Σας καλωσορίζω όλους. Στην ε, πρώτη από τις τέσσερις ε, συνεδρίες που έχουμε αυτή τη βδομάδα έχουμε φορτωμένη ημερησία διάταξη, μάλλον τρεις συνεδρίες θα έχουμε, τέσσερις γιατί έχουμε και μία ειδική συνεδρίαση για κλεισμένο το θυρών την πέμπτη το απόγευμα. Έχετε λάβει ήδη την ημερησία διάταξη. Μπορώ να σας ζητήσω να εγκρίνετε την ημερησία διάταξη. Πολύ ωραία εγκρίθηκε για τι ανακοινώσει του Προέδρου. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η συνεδρίαση είναι web streamed ε, γιατί είχαμε το πρώτο τμήμα για κλεισμένο των θηρών, ενώ τώρα ε, αναμεταδόμαστε και στο διαδίκτυο. Καλώς ορίζω όσους μας ακούνε και επίσης ε, έχουμε και την ε, επιστολή, το newsletter που καλύπτει την ημερησία διάταξη αλλά και κάποια άλλα θέματα. Αν θέλετε να λαμβάνετε αυτό το newsletter, μπορείτε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα. Βλέπετε τη διεύθυνση στο πίσω σελίδα. Και μπορώ να σας πω ότι έχουμε τώρα πάνω από χίλιου συγγεγραμμένους. Έτσι λοιπόν να πιέσουμε για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και τώρα των 2.000 το συντομότερο. Λοιπόν, έχετε τα πρακτικά από τις ε, συνεδριάσεις της 8ης Νοεμβρίου, 22 Νοεμβρίου και 9 Δεκεμβρίου. Αν υπάρχουν σχόλια για τα πρακτικά αυτά, παρακαλώ να τα διαβιβάσετε στη γραμματεία. Πριν από το τέλος της συνεδρίασης, αύριο το μεσημέρι θα τα λάβουμε τότε υπόψη. Διαφορετικά θα εγκριθούν τα πρακτικά όσα έχουν. Προχωρούμε λοιπόν τώρα στο ουσιαστικό θέμα της μερικής διάταξης για σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ που θα καλωσορίσω τον κύριο Μάντερς, ο οποίος είναι μέλος αυτής της Επιτροπής από το 2004, σίγουρα είστε φίλος του ΣΥΜΚΟ. Και θα περάσουμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση ε, των ονομάτων των κλωστοφοντουργικών προϊόντων και της σχετικής επισήμανσης των προϊόντων αυτών. Έχουμε εδώ ε, την κυρία Σελβίνη, την κυρία Σβένσον ε, και άλλους συναδέλφους που γνωρίζουν πολύ καλά αυτό το φάκελο. Και έχουμε και εκπροσώπους της Κομισιόν. Δεν ξέρω ποιος θα μιλήσει από την Κομισιόν. Κύριο Ζηράν. Μάλιστα, εσείς θα σχολιάσετε εκ μέρους της Κομισιόν. Να σας υπενθυμίσω ότι κάναμε την πρώτη ανάγνωση το 2009-2010 και τώρα έχουμε μία θέση του Συμβουλίου και θα μας πει και ο κύριος Μάντερς πώς την αξιολογεί. Έχουμε την κοινή θέση λοιπόν. Παρακαλώ κύριε Μάντερς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σωστή σύνοψή σας. Ε, έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωση και όπως ε, ξέρετε είχαμε συνδυασμό τριών υφιστάμενων ε, οδηγιών και τελικά η, προ... Κομισιόν πρότεινε κάτι ως κανονισμό και ξέρετε ότι ε, μου άρεσε εμένα γιατί τελικά έχουμε μια συνολική εισαγωγή νομοθεσία στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή έχουμε επικοδομητική συνεργασία με τους κοιόντις εισηγητές. Είχαμε μια συνεδρίαση άτυπου χαρακτήρα πριν από σήμερα. Όλοι περιβρίσκονταν, εγώ ήμουν πολύ ευτυχής και συζητήσαμε την προσέγγισή μας επίσης με την Κομισιόν. Είχαμε επικοδομητικές συνεδριάσεις και νομίζω ότι και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο είναι στο ίδιο μικρό πάνω κάτω. Αλλά ορισμένες φορές συμβαίνει σε εκθέσεις συναπόφασης στο Συμβούλιο ναι, μην ε, είναι διαθέσιμο να έρθει πιο κοντά στο Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή. Προσπάθησε η Βελγική Προεδρία, αλλά δεν τα κατάφερε στο θέμα αυτό. Αλλά ελπίζω ότι η Ουγγρική Προεδρία θα τα καταφέρει. Υπάρχουν ορισμένα επίμαχα ζητήματα, όπως ε, το θέμα της ε, σήμανσης της προέλευσης. Πρώτα είχαμε ένα διπλό σύστημα, υποχρεωτικό σύστημα για τα εισαγόμενα αγαθά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είχαμε και πάρα πολλές άλλες περιοχές, Καναδάς, Μεξικό, Ηνωμένε Πολιτείες, Βραζιλία, Αυστραλία, Ινδία, Κίνα, όλοι ζήτησαν το ίδιο από τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και γιατί να μην δημιουργήσουμε ίσως κανόνες και κατόπιν είχαμε και ένα εκούσιο σύστημα, αυτό είναι εκούσιο, ήταν σαφές, αλλά το Συμβούλιο φέρνει αντιρρήσεις και για τα δύο συστήματα και ούτε καν προτείνει κάποια λύση. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε και να προσπαθήσω να πείσω τους υπουργού μου για να μπλοκάρουν αυτά τα ζητήματα. Από τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε συναπόφαση σε περισσότερους τομείς και σε αυτό εδώ, εδώ βασιζόμαστε σε αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Δεν μπορούμε να συγχύζουμε τους καταναλωτές. Και σε αυτή την οδηγία μπορούμε να αποφύγουμε τη σύγχυση των καταναλωτών. Έχουμε μαζική υποστήριξη στο Κοινοβούλιο. Είχαμε και προηγουμένως την εκθέση μου και είχαμε και ευρία πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Αλλά υπάρχει εμπλοκή στην Κομισιόν επίσης. Σε σχέση με την ένδειξη της χώρας προέλευσης. Στην Ευρώπη δεν μπορούμε να έχουμε διακρίσεις μεταξύ των κρατών. Το Made in EU θα πρέπει να αναγράφεται για όλους. Επίσης, ένα λογοπήμαχο σημείο ήταν η γλώσσα ε, και τα σύμβολα για τα υφάσματα, για τα κλωστοφαντουργικά προϊόντα. Και πριν λίγες μέρες ε, βρέθηκε στο διαδίκτυο από τη συνάδελφο μία λίστα, ένας κατάλογος με την πρότασή μας ήδη και περίεργο που δεν τη δέχεται το Συμβούλιο. Πολλά έχουν ήδη επινοηθεί, πολλές φορές δεν το γνωρίζουμε και είναι κρίμα. Αν ενδιαφερόνται οι συνάδελφοι, έχω κάποια αντίτυπα και μπορώ να τους τα μοιράσω. Απλώς ε, θέλω να σας δείξω ότι αυτά τα πράγματα υφίστανται ήδη. Έτσι λοιπόν, γιατί να μην εξυπηρετήσουμε τους καταναλωτές και τη βιομηχανία και να τα δεκτούμε αυτά. Έχουμε επίσης ε, και άλλη επισήμανση για τα παιχνίδια. Εμείς ε, είπαμε ότι δεν είναι αυτό ειδικό ε, συγκεκριμένο πρόβλημα γιατί έχουμε την οδηγία για τα παιχνίδια. Είναι μια αυστηρή οδηγία. Τα υλικά που προέρχονται από ζώα, animal derived materials. Εδώ είχαμε προβλήματα, κυρίως το Συμβούλιο αντιτίθεται. Επίσης είδα ένα σχέδιο χρονοδιαγράμματος για να ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος, αλλά η μία συνεδρία προβλέπεται στο Στρασβούργο και νομίζω ότι πρέπει να αποφύγουμε να έχουμε πολλές ε, συναντήσεις στο Στρασβούργο. Ίσως μπορούμε να το τροποποιήσουμε λοιπόν κάπως αυτό το χρονοδιάγραμμα, αυτό το πρόγραμμα. Αλλά φυσικά είναι ανοιχτή πόρτα γιατί τώρα ξεκινάμε τη δεύτερη ανάγνωση. Δεν μπορούμε να θέσουμε νέα ζητήματα μπορούμε απλώ να ακολουθήσουμε το πνεύμα των τροπολογιών που έχουμε υιοθετήσει κατά την πρώτη ανάγνωση. Έτσι έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ε, ήδη έχω στείλει κάποιες επιστολές στους υπουργούς για να τους συναντήσω και να προσπαθήσω να τους πείσω. Και σε σχέση με την, το δίπλωμα της μπορούμε και να κάνουμε κάποια ανταλλαγή με τις υπουργού, γιατί κάποιες χώρες είναι αντίθετε ε, στο Ευρωπαϊκό Δίπλωμα της ενώ κάποιες άλλες ε, θέλουν να υιοθετηθεί και θέλουν να βρεθεί λύση. Έτσι λοιπόν, ε, αυτό δεν έχει να κάνει ειδικά με αυτό το ζήτημα, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, γνώση των Ευρωπαίων καταναλωτών σχετικά με την ενιαία αγορά. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει κάποιο κενό εδώ. Δεν ξέρουν οι καταναλωτές τι κάνει η ενιαία αγορά για αυτούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ γιατί κάνατε παρατηρήσεις που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο επίπεδο συνήθως και ε, καταλαβαίνετε επίσης ότι ε, στα πλαίσια της νέας νομοθεσίας για την ενιαία πράξη στην εσωτερική αγορά θα μπορούν να συμπεριληφθούν και τα όσα είπατε τώρα στο τέλος για την πληροφόρηση των καταναλωτών και ο αρμόδιος εισηγητής μας σαφώς θα μπορούσε να τις συμπεριλάβει τις παρατηρήσεις αυτές. Ως προς το συγκεκριμένο μου ζήτημα πρέπει να σας πω ότι έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Βρισκόμαστε στη δεύτερη ανάγνωση πιέζουν οι διορίες και καλείστε να στείλετε στις 8 Φεβρουαρίου το τελικό κείμενό σας, το οποίο πρέπει να πάει για τη μετάφραση, δηλαδή το σχέδιο συστάσεων που θα κάνετε. Στις 28 Φεβρουαρίου θα συζητήσουμε το κείμενο αυτό και η Δευτέρα Μαρτίου είναι η ημερομηνία η τελική για την κατάθεση τροπολογιών και στι 22 Μαρτίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Στη συνέχεια βέβαια οι οποιασδήποτε διαπραγματεύσει θα έχουν να κάνουν με την βούληση των ίδιων των συντονιστών να περάσουν σε περαιτέρω διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο για να καταλήξουν σε μία συμφωνία πριν την ψηφοφορία τη δεύτερη ανάγνωση. Και βέβαια αυτό να εξαρτάται από εσά και από του συντονιστέ. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα είπατε. Μολονότι το Συμβούλιο έχει δεχθεί αρκετέ από τι τροπολογίε μα, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια ουσιαστικά ζητήματα ακόμα για τα οποία δεν έχουμε συμφωνήσει. Πράγμα το οποίο κάνει, θα έλεγα, την δική σας την εργασία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και θα απαιτηθούν πολλές επαφές μεταξύ ημών και του Συμβουλίου. Και σαφώς βέβαια καλωσορίζουμε και την Ουγγρική Προεδρία καθώς επίσης και τον αρμόδιο της, την κυρία Γιάκο μάλλον, την αρμόδια της Ομάδας Εργασίας Συμβουλίου. Ας ακούσουμε τώρα τι έχουν να πούνε οι σκιώδεις ηγητές. Κυρία Κόμπη πρώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την εξαιρετική δουλειά του κυρίου Μάντερς ε, και όλων των άλλων των σκιώδων εισηγητών. Προσπάθησαν να βρουν ε, μια κοινή σκοπιά, γιατί ήδη ευρύναμε τις ε, θεματικές που αποκλείονταν αρχικά από αυτόν τον κανονισμό, αλλά θεωρούμε ότι η διεύρυνση οφειλόταν στο ότι εντάχθηκε η ε, καταγωγή, η σήμανση της καταγωγής και όλα αυτά ε, έχουν να κάνουν με την καλύτερη προστασία του καταναλωτή. Στις 18 Μαρτίου είχαμε μια ψηφοφορία στο Κοινοβουλίο και αυτό αποτελεί ένα βήμα προς τα μπρος γιατί είχαμε ευρεία πλειοψηφία από όλες τις πολιτικές ομάδες. Και φυσικά πρέπει τώρα να αντιπαραταχθούμε με το Συμβούλιο, που το οποίο δεν έχει εκφράσει καμία θέση σε σχέση με την ένδειξη καταγωγή. αν και πέντε κράτη-μέλη δήλωσαν την πλήρη υποστήριξή τους και ε, δεν μιλάμε μόνο για χώρες μικρές, γιατί μιλάμε για Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Λιθουανία. Εγώ θεωρώ ότι ο σκοπός της ε, ονομασίας καταγωγής ε, που συζητήθηκε και στο φάκελο Μοσκαντινή είναι και σε αυτή την περίπτωση ε, το στοιχείο που συζητήθηκε περισσότερο και έχει δύο στόχους. Καταρχήν να ενισχύσει την προστασία των καταναλωτών γιατί ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει απόλυτα πλήρως ε, που κατασκευάζεται το προϊόν και μόνο το τελευταίο ε, στοιχείο, το τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας ε, δείχνει την τοποθεσία κατασκευής και είναι αν αναγράφεται μόνο αυτό τότε δεν δείχνει που έχει κατασκευαστεί το προϊόν. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, αν γράφουμε ότι έχει φτιαχτεί στην Ιταλία, στη Γαλλία και προσθέτουν έχουν προσθεθεί τα κουμπιά ε, στο ρούχο, δεν νομίζω ότι ε, καλύπτουμε την ε, τοποθεσία κατασκευή του προϊόντο. Επίση, έχουμε μία σειρά επιχειρήσεων που έχουν μεταφέρει τι εγκαταστάσει του και. εγώ θεωρώ ότι ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πιο σημαντικό μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό και το Συμβούλιο να το λάβει αυτό υπόψη και η νέα Ουγγρική Προεδρία. Γιατί θα μπορούσε η νέα Ουγγρική Προεδρία να οδηγήσει σε εξαιρετικά αποτελέσματα, καθώ αυτά τα αποτελέσματα ζητούνται και από του καταναλωτέ για να γνωρίζουν καλύτερα ε, τι αγοράζουν και από πού προέρχονται οι αγορέ του. Ε, από το 2005 έχει μπλοκαριστεί αυτό το θέμα από το Συμβούλιο. Ίσως ε, ήρθε η στιγμή να απελευθερώσουμε, να απεμπλοκάρουμε την κατάσταση τώρα. Ε, και επίσης ε, θεωρώ ότι η βούληση αυτής της Επιτροπής είναι να ενισχύσει την ενιαία αγορά. Και με το φάκελο Μόντι ε, αυτό το στόχο έχουμε θέσει. Και ένας ακόμη στόχος είναι να ενισχύσουμε τις εσωτερικές οικονομίες τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή. Και καθώς ο τομέας των κλωτοφεστουργικών είναι ένας από τους κύριους τομείς μαζί με τον τουρισμό που αποτελείται με μηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας, νομίζω ότι εδώ μιλάμε για ένα ε, κύριο τομέα που πρέπει να προστατεύσουμε. Και γι' αυτό το λόγο εγώ συμφωνώ και με όλα τα υπόλοιπα σημεία που υπογράμμισε ο εισηγητή και τον υποστηρίζω πλήρως. Θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο ο κύριος Μάντερς ε, να συνεχίσει να υποστηρίζει τους κανόνες για την ε, σήμανση καταγωγής ε, γιατί δύο φορές είχαμε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου και για τα κλωστοβδουργικά και για το φάκελο Μοσκαρδίνη. Έτσι λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στον κύριο Μάντερς θα έχει την πλήρη υποστήριξη και από μένα και από την ομάδα μου. Uh, thank Σας ευχαριστούμε κυρία Κόμη, η κυρία Σαλαμόζα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Μάντερς για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. αποφασιστική σημασία για μας κατά τη δεύτερη αυτή ανάγνωση είναι να φροντίσουμε οι καταναλωτές τελικά να λαμβάνουν καλύτερες και σαφέστερες ε, πληροφορίες σχετικά με τα ε, προϊόντα υφασμάτων που αγοράζουν. Αυτό είναι το δικό μας μήνυμα και γι' αυτό θα πρέπει να αγωνιστούμε διότι φαίνεται ότι το Συμβούλιο δεν είναι διατεθειμένο να μας ε, το δώσουν αυτό διότι έχουν ε, υποχωρήσει όσον αφορά κάποιες από τις τεχνικές ε, απαιτήσεις τους, ε, όχι όμως όσον αφορά τις προτάσεις μας που διευκολύνει τον καταναλωτή να γνωρίζει τι είναι αυτό που αγοράζει. Γι' αυτό συμφωνώ με τον Πρόεδρο ότι διαφωνούμε στα επί και θα πρέπει το Συμβούλιο να υποχωρήσει για να πετύχουμε ε, μια καλή συμφωνία. Είμαστε διατεθειμένοι να ε, διαπραγματευτούμε, αλλά θα πρέπει ε, να υποχωρήσουν κάπως. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Μάντες για την πολύ καλή δουλειά που κάνει και για την συνεχή ενημέρωση που μας κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Σας ευχαριστούμε κυρία Σαλτεμόζη, κυρία Ρούλη. Μπορώ να είμαι σύντομη. Ο κύριος ε, Μάντερς ε, θα καταβάλει προσπάθειες, αλλά εγώ από την αρχή ήμουν σκεπτική σχετικά με το αν το Συμβούλιο σε ένα τεχνικό θέμα ε, θα είναι διατεθειμένο να συμπεριλάβει και τα πολιτικά μας αιτήματα. Να δούμε τι θα πετύχουμε στη δεύτερη ανάγνωση. Η κυρία Μακλάκη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να θυμηθούμε όλοι ότι ο στόχος του κανονισμού αυτού ήταν να διευκολυνθεί η εισαγωγή νέων υφασμάτων στην αγορά και να απλοποιηθεί η, η επισήμανση. Ε, οτιδήποτε λοιπόν έχει να κάνει με την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ε, του κανονισμού αυτού είναι ενάντια στην αρχική μας πρόθεση. Ε, θα πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποιες προσαρμογές στο, ε, στα σημεία αυτά. Όσον αφορά την ε, σήμανση προέλευσης, ε, να δούμε τι θα μπορούμε να πετύχουμε, μήπως θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα ε, προαιρετικό σύστημα. Και όσον αφορά την ε, ρήτρα αναθεώρησης που περιλαμβάνει πολλά από τα πολιτικά ζητήματα, ήταν αρκετά αναλυτική και ε, περιείχε υπερβολικές απαιτήσει. Πιστεύω θα πρέπει να συζητήσουμε τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η ρήτρα αυτή αναθεώρησης, αν τη θέλουμε. Ε, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να περιέχει σημεία που να ε, περιέχουν προσθέμενη αξία για τον καταναλωτή. Να φροντίσουμε να υποστηρίζουμε τις ε, μικρές επιχειρήσεις, τους μεμονωμένους ράφτες Ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε περιθώρια λιγμού, να συμπεριλάβουμε κάποιες από τις προτάσεις της Κομισιόν, ώστε να πετύχουμε αποτελέσματα τώρα προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Ε, λυπάμαι που σας ε, τα χαλάω, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτές τις πληροφορίες αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Όχι, νομίζω ότι και εσείς και η κυρία Ρούλε. Ε, είπατε αυτό που ήθελα να θυμίσω στην Επιτροπή μας ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι όσον αφορά την νομοθεσία αυτή. Είμαι βέβαιος ότι η Κομισιόν θα μας το θυμίσει αυτό. Ε, το κατά πόσο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ε, την νομοθεσία αυτή πολιτικά για να πετύχουμε άλλου στόχου, ε, αυτό θα το αποφασίσει η Επιτροπή. Αλλά όσον αφορά την σήμανση προέλευση, αυτό είναι θέμα εμπορικό. Και ακόμα και αν θέλαμε δεν θα μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε στην πρόταση αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι οι σκιώδεις συζητητέ θα πρέπει να συζητήσουν ποιοι είναι οι πολιτικοί τους στόχοι και ποιοι είναι οι κατάλληλοι τρόποι να τους πετύχουν μήπως θα μπορούσαμε να πετύχουμε μία δήλωση της Κομισιόν σχετικά με πρόσθετες εργασίες ε, που πρέπει να γίνουν, ε, κάτι που να μην συμπεριλαμβάνεται στη βασική νομοθεσία. Ξέρουμε ότι είχαμε επιτυχία σε κάποιες περιπτώσεις όπου η Κομισιόν δέχτηκε σαφείς προθεσμίες ε, σχετικά με τις μελλοντικέ εργασίες. Είμαι βέβαιος ότι ο εισηγητής θα το έχει αυτό κατά νου να δω ε, εάν υπάρχει άλλος από την Επιτροπή μας που θέλει να πάρει το λόγο, διότι ακούσαμε όλου του κοιόδες Συγητέ. Εάν όχι, να ζητήσω από τον κύριο Ζηράου από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ε, πει πω πιστεύει ότι θα προχωρήσει το θέμα αυτό. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να επαναλάβω τα όσα άλλωστε είχε πει στην τελευταία της ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιδρώντας τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να πω δηλαδή ποια είναι τα πια ουσιαστικά σημεία για μας. Ουσιαστικά αυτά που έχουν να κάνουν με την τροπολογία 19 εξαιρέσεις για τα καταπαραγγελία προϊόντα το να χρησιμοποιούνται επίσης συγκεκριμένα σύμβολα όσον αφορά τη σήμαση των προϊόντων και επίσης τι μπορεί να γίνει με τα παιχνίδια εκείνα τα οποία είναι φτιαγμένα από υφάνσιμες σύνες, από υφάσματα. Θα μπορούσαμε σε κάποια άλλα σημεία να εξετάσουμε κάπως και τη διατύπωση. Ουσιαστικά όμως έχουμε τροπολογίες που γίνονται αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί της αρχής, δηλαδή μπορούμε να τις ε, δεχθούμε. Γνωρίζουμε όμως ότι οι τροπολογίες εκείνες που έχουν να κάνουν με την χώρα προέλευσης και οι τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τα υλικά ζωικής προέλευσης είναι τροπολογίες αρκετά φιλεγόμενες στο Συμβούλιο, αρκετά επίμαχες. Έχουν υποστηριχθεί όμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τον κανονισμό αυτό. Και αυτό γιατί πιστεύουμε ότι το να καταφέρουμε να αντικαταστήσουμε τις τρεις οδηγίες με έναν κανονισμό είναι ουσιαστικά ένα εγχείρημα το οποίο θα ωφελήσει τόσο τις εθνικές αρχές όσο και τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Τζιράου. Και όπως ε, σας είπα, χαιρετήσαμε μάλλον και την ε, Ουγγρική Προεδρία. Θα έχουμε τη δυνατότητα να του ακούσουμε και στο μέλλον. Δεν ξέρω αν ο συγητή ο κύριος Μάντερ θέλει να πει κάποια πράγματα περισσότερο, αν έχει να πει κάτι για το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει ήδη ένα χρονοδιάγραμμα, το αναφέρατε όμω εσεί εσεί Πρόεδρε, δεν υπάρχει λόγο να επαναλάβουμε αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι όλα σαφή. Έχω μπροστά μου το χρονοδιάγραμμα, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Θα ήθελα όμω να πω ότι θα ήθελα να συνεργαστώ, όπω άλλωστε είπαν και οι συνάδελφοι, και ελπίζω ότι στα τέλη Μαρτίου θα καταφέρουμε να βρούμε μια λύση, όταν θα χρειαστεί να ψηφίσουμε δηλαδή κιόλα και καταλαβαίνετε ότι πρέπει και οι τρεις να συνεργαστούμε, δηλαδή και τα τρία θεσμικά όργανα και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε με την ε, απαραίτητη βούληση να, τα καταλήξουμε συμφωνία. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Πρωτού προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να πω ότι εφόσον εδώ ο κύριο Μάντερ, ότι ε, στην πρώτη σελίδα του ενημερωτικού μα φυλαδίου αναφερόμαστε πλέον ε, στα κοινά στάνταρτ, στα κοινά πρότυπα κινητή τηλεφωνία ε, και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και εσά κύριε Μάντερ για την εργασία που κάνατε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία προκειμένου να καταλήξουμε στο νομοθέτημα αυτό. Και η κυρία Ρούλ επίση ήταν η συγγήτρια για το ζήτημα αυτό. Θα ήθελα και να την ευχαριστήσω, μόλι ότι δεν με ακούει αυτή τη στιγμή. Χάιντι. Ναι, το ζήτημα αυτό θα πρέπει να σας απασχολήσει και τώρα, εφόσον αναφερόμαστε και στα tablets. Πάντως, λέει ο Πρόεδρος, μετά την πάρα πολύ καλή έκθεση που υπήρχε για την πολιτική συμβάσεων, δημοσίων συμβάσεων, την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιοποίηση μια πράσινη δίβλο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Πολιτική Δημοσίων Συμβάσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, μπορείτε να αντιδράσετε και ω προ αυτό και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό και να θεωρήσει πολλέ πτυχέ τη πολιτική δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο κύριος Μάντερς. Σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε τώρα ότι όσον αφορά τις, τα πρότυπα στα οποία αναφερθήκατε. Αν καταφέρουμε να συνεργαστούμε καλά, θα καταφέρουμε να πετύχουμε παγκόσμια πρότυπα πλέον, όχι μόνο πρότυπα τα οποία θα έχουν να κάνουν με την πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Πρέπει τώρα να προχωρήσουμε σε ένα άλλο σημείο το οποίο έχει παγκόσμιο αντίκτυπο και αυτό. Αναφέρομαι στην ανθερημένη πρόταση για την έγκριση τύπου και εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων. Ο κύριος Βάντε Κάπα είναι ο συγητής μας, ο οποίος εργάστηκε πολύ σκληρά για το ζήτημα αυτό. Θα μας πει σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει και έχουμε και τους σκιώδεις εισηγητές μας, Μάντερς, Ρούλε, εγώ ίδιος για την δική μου την πολιτική ομάδα και ο κύριος Σαλβίνη, καθώς επίσης και άλλοι. Υπάρχουν πολλοί σκιώδη συγητοί για το ζήτημα αυτό. Το λόγο έχει καταρχά ο κύριο Βάντεν Κάπ για να μα πει πώ προχωράμε με το ζήτημα αυτό. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τώρα είναι η σειρά μου. Μετά τον κύριο Μέντες. Από τις 30 Νοεμβρίου του 2010 είχαμε πάρα πολλή δουλειά. Στις 30 Νοεμβρίου είχαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Και από τότε μίλησα με ομάδες ενδιαφέροντος και με τη βιομηχανία και με τον τομέα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την όλους για την υποστήριξη που έλαβα σε αυτό το project. Και έχουμε προγραμματίσει και τρεις επισκέψεις ε, για το Φεβρουάριο. Έχω προετοιμάσει μία σειρά ερωτήσεων. Έχω ήδη διαβιβάσει αυτές τις ερωτήσεις στους κοιόδης συζητητές και ελπίζω ότι σήμερα ή τις επόμενες εβδομάδες θα λάβω απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Θα μπορέσω να απαντήσω στις ερωτήσεις αυτές που ε, έχουμε βάλει στον κατάλογο. Ποια είναι τα κυρία σημεία. Η συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί σε τέσσερις κυρίους τομείς. Καταρχήν, τι πρέπει ή τι δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στον κανονισμό. Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες πτυχές που δεν είναι ιδιαίτερα σαφείς για τα οχήματα, τα ηλεκτρικά και επίσης εμείς δεν θέλουμε καθόλου να μπλοκάρουμε την καινοτομία και την πρόοδο. Δεύτερο θέμα, τα μέτρα ασφαλείας γιατί προτείνονται νέα μέτρα ασφαλείας ε, τα οποία είναι αρκετά αυστηρά αλλά τελικά μπορούμε να ρωτηθούμε μήπως αυτά μέτρα ασφαλείας κοστίζουν περισσότερο από το ίδιο το όχημα και έτσι λοιπόν ε, και εδώ θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Επίσης, συζητείται και η δυνατότητα της προσαρμογής. Ένα ακόμα στοιχείο είναι τα περιβαλλοντικά μέτρα. Πολλές φορές ε, η βιομηχανία θέλει να προχωρήσει γρήγορα, εντάξει, μπορεί να προχωρήσει αν θέλει να εισαγάγει και μέτρα που να φορούν το περιβάλλον. Κατόπιν ε, έχουμε και τα διάφορα πληροφορίες ε, για τα οχήματα προς επισκεφτή δεν πρέπει να στέλνετε μόνο στους αντιπροσώπους, αλλά και στους χρήστες ε, αυτών των ε, οχημάτων, αλλά και στα συνεργεία. Αυτή είναι η δική μας θέση. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βέστφαλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Είναι ιδιαίτερα τεχνικό το ζήτημα. Ε, και έτσι περνάω στον αρκετά μακρύ κατάλογο των ερωτήσεων μου. Βρισκόμαστε στην αρχή των εργασιών ε, κάποιες ε, επισκέψεις θα γίνουν όπου θα απαντηθούν κάποια από τα θέματα αυτά, αλλά ε, να κάνω κάποιες προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να προστατεύσουμε όσο μπορούμε τους οδηγούς μηχανοκίνητων οχημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο μειώνονται τα θύματα τροχαίων, αλλά ιδιαίτερα όσον αφορά τα τα μηχανάκια, ε, ε, τα δίκυκλα, ε, παραμένει πολύ υψηλός ο βαθμός των θυμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να παρέχουμε όσο γίνεται καλύτερη προστασία των οδηγών μοτοσυκλετών. Η διαδικασία θα είναι αρκετά μακρά. Θα πρέπει να απαντηθούν ε, κάποια ερωτήματα. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι εγώ όταν μιλάω για συστήματα ABS εννοώ το σύστημα anti-blocking διότι υπάρχουν ε, διαφορετικές μεταφράσεις και ερμηνείες του όρου. Εγώ πιστεύω ότι κάποια ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν είναι είναι τεχνικά εφικτό ε, τα ε, οχήματα ε, των κατηγοριών L1, L2, δηλαδή τα μικρά μηχανάκια και τα τρίκυκλα, αν είναι δυνατόν αυτά να έχουν σύστημα ABS. Δεύτερον, τι δυσκολίες θα έχουν η παραγωγή μικρών σειρών οχήματων, τι δυσκολίε θα έχουν οι παραγωγοί αυτοί εάν γίνει μια τέτοια τροποποίηση των ε, κανόνων. Επίσης, συνδυασμένα συστήματα φρένων, τα CBS ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο με τα ε, ABS. Και τελευταία ερώτηση. Το ABS, εάν παρέχει περισσότερη ασφάλεια από το CBS, δεν θα πρέπει τότε στον κανονισμό σαφώς να το αναφέρουμε αυτό και να καταστήσουμε υποχρεωτικό το ABS. Αυτές είναι κάποιες βασικές ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντηθούν. Είμαι βέβαιη ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα βρούμε απαντήσεις. Θα ήθελα να κλείσω εδώ και προσβλέπω στη συνέχιση της καλής συνεργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βέστφαλ που θέσατε τα βασικά ερωτήματα της πρότασης αυτής η κυρία Ρούιλε. Όχι, συγγνώμη, ο κύριος Μάντερς. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τον κύριο Βεντεκάμπ. Ε, είναι πολύ μετριόφρον. Εν τω μεταξύ έχουμε γίνει φίλοι και τελευταία συνεργαζόμαστε. Μπορώ να σας πω ότι ο συνάδελφος είναι και πολύ καλός ε, μοτοσυκλετιστής. Τώρα έχουμε αυτή την πολύπλοκη νομοθεσία σε σχέση με την έγκριση ε, τύπου των ε, οχημάτων κατηγορία Ελλήνα, ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστημα και θέλουμε να το καταστήσουμε σαφέστερο και απλούστερο. Εξ ονόματο τη ομάδα των φιλελευθέρων, σκεφτόμαστε ότι οι περιβαλλοντικές προϋποθέσεις στην Ευρώπη πρέπει να τυποποιηθούν έτσι ώστε να έχουμε μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για μένα το πιο σημαντικό είναι το θέμα της ασφάλειας για τα οχήματα τρίκυκλα και τετράκυκλα αν ένα τέτοιο όχημα δεν είναι ασφαλές τότε είναι πολύ πιθανό να συμβεί ατύχημα πριν ε, κάποια χρόνια εμένα δεν με είδε ένα αυτοκινητιστής και ε, πολύ συχνά όσοι οδηγούν αυτοκίνητα δεν βλέπουν ε, αυτούς που οδηγούν μοτοσικλέτες γιατί δυστυχώς δεν προσέχουν τα πιο μικρά οχήματα και μιλώ και για ποδήλατα, μοτοσικλέτες κτλ. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα εργάζεται επί του θέματος της ασφάλειας και προβλέπει να εισαγωγεί διάφορα μέτρα ασφαλείας. Ελπίζουμε αυτό να καταλήξει σε ένα αυτό αποτέλεσμα. Εμείς υποστηρίζουμε και την ιδέα να έχουμε ένα σύστημα ε, με φώτα που θα ανάβουν αυτόματα όταν ε, λειτουργεί το όχημα, γιατί κατά τέτοιο αυξάνει την ασφάλεια. Επίσης είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές ε, να μπορούν να λαμβάνουν την έγκριση για νέα είδη μηχανών κινητήρων. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε την κοινοτομία. Εδώ συμφωνώ με τον εισηγητή. Έτσι λοιπόν πρέπει να είναι δυνατόν να γίνουν κάποιε μικρέ προσαρμογέ και σε μετέπειτα στάδιο. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να ανταγωνιστεί και με τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί και αυτό είναι στόχο μα. Αυτά. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, οι συγητές και οι συγητές μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία, όλοι αγαπούν ε, τα οχήματα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και είναι την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει. Κυρία Ρούλα. Εγώ δεν είμαι μοτοσυκλετίστρια. Ε, ως, ε, όταν ήμουν παιδί Καθόμουν στη μηχανή, ε, ω παιδί καθόμουν στην μπανάνα ε, μέχρι να αποκτήσει η οικογένειά μου αυτοκίνητο. Ε, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για, την, για τις πολύ χρήσιμες ερωτήσεις και να ξεκινήσω από τις γενικές παρατηρήσεις. Αναφέρεσαι στις δαπάνες. Φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το κόστος. Υπάρχει όμως και εξωτερικό κόστος επιβάρυνση για το περιβάλλον, το θέμα της, ε, του, του περιορισμού των φυσικών πόρων, του πετρελαίου. Ε, θα πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη όταν μιλάμε για το κόστος ε, και όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και μπορεί να σκεφτεί κανείς τι σχέση έχει το πεδίο εφαρμογής με το περιβάλλον. Εγώ, βρίσκομαι, εγώ προέρχομαι από τη Στουτγάρδη χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερα ποδήλατα και μοτοποδήλατα. αυτά όμως δεν έχουν αποκλειστεί από την Κομισιόν από το πεδίο εφαρμογή. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα πρέπει να ε, αποκλείται από το πεδίο εφαρμογή ε, της νομοθεσίας αυτής, ε, διότι ε, τα ηλεκτρικά ποδήλατα ε, δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να αποκλειστούν. Έχουν ε, περιορισμό στην ταχύτητα και χρειάζονται διαφορετική μεταχείριση ώστε να επιτρέψουμε την καινοτομία και για να δώσουμε τη δυνατότητα σε ηλικιωμένους να ε, χρησιμοποιούν ηλεκτρικά ποδήλατα. Δεν έχει νόημα ε, ξαφνικά να τους βλέπουμε με κράνος ε, να τριγενάνει στη γειτονιά. Έτσι δεν θα χρησιμοποιήσουν ποτέ ηλεκτρικά ποδήλατα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε επικόντως με το θέμα αυτό. Όσον αφορά την επιβάρυνση για το περιβάλλον, τρίτο θέμα, θα ήθελα να πω ότι ο σχετικός τομέα ήδη λέει ότι είναι πολύ πιο εύκολη η μετατροπή και η μετάβαση ε, ε, στα οχήματα αυτά δεν έχει νόημα να καθυστερούμε. Θα πρέπει και εδώ στην Ευρώπη να δώσουμε το καλό παράδειγμα ώστε και σε αναπτυσσόμενες χώρες να δώσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται πιο φιλικά προς το περιβάλλον ε, μηχανοκίνητα ε, δίκυκλα Ε, χρήσιμο θα είναι όσον αφορά την τεχνολογία να είμαστε καινοτόμοι. Ε, θα πρέπει και η πολιτική να ε, προσαρμοστεί αναλόγως. Όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να τα συζητήσουμε εντελεχώς, αλλά όσον αφορά το κόστος θα ήθελα να πω κάτι γιατί αναφέρθηκε. Εάν δεν είναι υποχρεωτικό υποχρεωτικές ε, κάποιες ε, παροχές ε, τότε θα είναι και πιο ακριβές από το εάν παρέχονται αυτομάτως με το όχημα όπως για παράδειγμα τα ABS. Επίσης είναι πολύ σημαντικό και επίγον να ασχοληθούμε με την αγορά επισκευών να υπάρχουν ε, να υπάρχει σωστή πρόσβαση σε πληροφορίες. Είναι πολύ σωστές οι ερωτήσεις σας ε, και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λίγα λόγια από μένα στην ιδιότητά μου ως σκιώδη εισηγητή, διότι νομίζω ότι οι συνάδελφοι εντόπισαν κάποια ζητήματα. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Βαντεκάμπ Καταρχήν επειδή επιδιώκει μια μεθοδική και χρήσιμη προσέγγιση στο θέμα και που μας δίνει ε, τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με εμπειρογνώμονες για το θέμα αυτό, διότι μιλάμε για ε, την κρίση του νομοθέτη και των ε, τεχνικών εμπειρογνωμόνων και τελικά θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση και να δούμε αν συμφωνούμε με τη θέση της Κομισιόν. Καταρχήν είναι σημαντικό να μην σκεφτόμαστε τα μηχανάκια με τον ίδιο τρόπο που σκεφτόμαστε τα αυτοκίνητα. Έχει πολύ ευρύ πεδίο εφαρμογή ε, ο κανονισμός αυτό. Σε κάποιες... Ε, ε, πτυχές ε, άπτονται και των ηλεκτρικών ποδηλάτων, ε, των οποίων η τεχνολογία όμως προέρχεται από το κανονικό ποδήλατο και όχι από, το, και όχι από τα μηχανάκια. Σε κάποιες πόλεις ο, ο κόσμος ενθαρρύνεται να αγοράσει την νέα γενιά μικρών μηχανοκίνητων οχημάτων που είναι σαν σκούτερ. Το θέμα των ε, μηχανικών λύσεων, το κόστος τους, ε, το, ε, τα ωφέλη τους, η συζήτηση αυτή είναι πολύ σημαντική και νομίζω ότι υπάρχει συνένεση ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά τα ABS για τα ακριβά μηχανάκια που ε, ε, βλέπονται για μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων, για τα μικρά μοτοποδήλατα δεν ε, θα προβλέπετε κάτι τέτοιο μάλλον, διότι ε, ούτε αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, ούτε ταξιδεύουν σε μεγάλες ε, αποστάσεις. Θα πρέπει όμως να ασχοληθούμε με τις ενδιάμεσες κατηγορίες. Υπάρχουν και κάποια ευρύτερα θέματα σχετικά με το κατά πόσο θα είναι αποτελεσματικά κάποια μέτρα. Όσοι γνωρίζουν την χρήση ABS στα αυτοκίνητα θα γνωρίζουν ότι ε, πολλοί οδηγοί κατά τη διάρκεια ατυχημάτων δεν φρέναραν αρκετά ώστε να, ε, να μπει σε λειτουργία το σύστημα EPS. Δεν ήξεραν ε, πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό και δεν το εμπιστεύτηκαν να φρενάρει το αυτοκίνητο. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα σύστημα που έλεγχε Electronic Assist System ώστε σε περίπτωση ανάγκης εάν φρενάρει κανείς δυνατά να τεθεί σε λειτουργία το anti-block system, το ABS. Ε, όσον αφορά τα μηχανάκια, είναι διαφορετική κατάσταση, διότι η σταθερότητα του οχήματο είναι τελείω διαφορετική ε, και θα πρέπει να ε, ρωτήσουμε του εμπειρογνώμονε εάν θα είναι αποτελεσματικό το σύστημα ABS, διότι οι οδηγοί δεν έχουν εμπειρία με τη χρήση του Θα πρέπει να βρούμε την πιο οικονομική και πιο αποτελεσματική λύση. Ε, ξέρω ότι κάποιοι από εσά θα επισκεφτείτε ένα κέντρο ελέγχων την Πέμπτη για να συζητήσετε τα θέματα αυτά. Όσον αφορά τι εκπομπέ, ε, αναφέρθηκαν και εδώ κάποια σημαντικά θέματα. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ε, θέματα παρέμβαση ε, στα οχήματα, τροποποίηση των οχημάτων, αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν μηχανάκια που τους αρέσει να τα τροποποιούν, να αλλάζουν διάφορα πράγματα. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, συστήματα επιβολής του νόμου για να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, εάν θέλουμε να είναι ε, χρήσιμη η νομοθεσία μας. Ε, και φτάνω στο τελευταίο θέμα που έχει να κάνει με την ασφάλεια. Η κυρία Βέσταλ αναφέρθηκε στα θύματα μεταξύ των μοτοσυκλετιστών. Ε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι τα θύματα εδώ δεν ε, έχουν να κάνουν μόνο με την τεχνολογία. Υπάρχει το θέμα της εκπαίδευσης των οδηγών, ε, το επίπεδο δεξιοτήτων, το οποίο έχει αντιμετωπιστεί εν μέρη τώρα με τις διάφορες κατηγορίες διπλωμάτων. Υπάρχει το θέμα των, του κράνους, αλλά νομίζω ότι η ασφάλεια το, για τους μοτοσυκλετιστές ε, ε, ε, έχει να κάνει και πολύ με τον σχεδιασμό των δρόμων και με την ορατότητα και με διάφορα εμπόδια που υπάρχουν στο δρόμο. Είναι λοιπόν πολύ πιο πολύπλοκο το θέμα αυτό είναι μεγάλη η ποικιλία των οχημάτων ε, που συζητάμε εδώ πέρα και νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε ε, μία ενιαία λύση αλλά να εξετάσουμε την ε, προσέγγιση κατά κατηγορίες της Επιτροπής. Χρήσιμο δηλαδή θα είναι να προτείνουμε κάποια πράγματα τα οποία να μην είναι αδύνατο να επιτευχθούν. Προσβλέπουμε λοιπόν στην ε, καλή συζήτηση για το θέμα αυτό. Υπάρχει κανείς άλλος ε, που να θέλει να λάβει το λόγο που να μην είναι σκιώδης εισηγητής. Η κυρία Ρόιτοβα, ο κύριος Μαρτίνη βλέπω ότι είναι εδώ, θα, τον, ε, θα δώσω το λόγο σε λίγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση σε όλους τους εισηγητές. Να εξτάσουν λίγο το ζήτημα των τεχνικών ελέγχων. Από όσο γνωρίζω, και δεν ξέρω αν κάνω λάθος ή όχι, γιατί δεν είναι ακριβώς ο δικός μου τομέας αυτός, από ό,τι φαίνεται όμως δεν υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση των τεχνικών ελέγχων που γίνονται στα αυτοκίνητα. Και συγκεκριμένα για τα οχήματα τα οποία εξετάζουμε σήμερα. Από ό,τι φαίνεται η κατάσταση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και από ό,τι φαίνεται είναι πολύ δύσκολο να καταφέρει κανείς να έχει τεχνικό έλεγχο στον ε, χώρο, στην χώρα εκείνη που είχε ταξινομηθεί το όχημα. Ουσιαστικά εγώ ακόμα και ζώντας εδώ πέρα στο Βέλγιο συναντώ πάρα πολλά προβλήματα όταν θέλω να κάνω τεχνικό έλεγχο στο αυτοκίνητό μου. Μου λένε πολύ συχνά ότι θα πρέπει να πάω στην χώρα που αγόρασα το αυτοκίνητο αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι και το ζήτημα τεχνικού ελέγχου θα πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά. Πρόεδρος. Κύριε Ρόιτερβερ, θεωρώ ότι υπάρχει ήδη μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα αυτό, για το τεχνικό έλεγχο δηλαδή των οχημάτων και οι συναδελφοί μας στην αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου εξετάζουν ήδη το ζήτημα αυτό. Καταλαβαίνετε ότι εμείς ε, δεν μπορούμε να βγούμε από τις αρμοδιότητες δικής μας Επιτροπής. Η Επιτροπή Μεταφορών ενδεχομένω να είναι πιο αρμόδια. Αν δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν το λόγο, δίνω το λόγο στον κύριο Μαρτίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Πολύ σύντομα θα ήθελα να σχολιάσω και εγώ να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή και τους σκιώδη εισηγητές για τις παρατηρήσεις τους. Θεωρώ ότι οι παρεμβάσεις παραβαν χώρα και που ακούσαμε σήμερα το πρωί πραγματικά αναφέρονται στα ουσιαστικά ζητήματα τα οποία διέπουν και τη δική μας εργασία και που θα χαρακτηρίσουν ουσιαστικά την εργασία που θα κάνουμε τους επόμενους μήνες. Όσον αφορά τώρα τα ζητήματα τα οποία ακούσαμε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Να επιβεβαιώσω καταρχάς ότι ε, όσον αφορά την πτυχή της ασφάλειας και ιδίω και όχι μόνο όσον αφορά το ζήτημα του ABS και τα συστήματα απέδησης, και εμείς πολύ προσεκτικά στην ε, ανάλυση αντικτύπου λάβουμε υπόψη μας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, καθώς επίσης και τα δεδομένα που έχουμε για τα ατυχήματα στην Ευρώπη. Σίγουρα τα δεδομένα αυτά δεν είναι εύκολο να τα αξιολογήσουμε, να τα αναλύσουμε ή και να τα συλλέξουμε ακόμα. Πάντως καταβάλαμε προσπάθειες προκειμένου να πετύχουμε την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην απόλυτη ανάγκη αύξησης του επίπεδου ασφάλειας στον τομέα αυτό και από την άλλη στο να έχουμε τον καλύτερο δυνατό θετικό αντίκτυπο για το κόστος και για τους καταναλωτές. Έχουμε λοιπόν κατά νου ότι τα μοτοποδήλατα, οι μοτοσυκλέτες στις αστικές κυρίως περιοχές σαφώς θα πρέπει να συμβάλλουν στο να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά θα πρέπει να συμβάλλουν και στη μείωση των εκπομπών και αναφέρομαι κυρίως βέβαια στις αστικές περιοχές. Σαφώς λοιπόν και τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το άλλο ζήτημα το οποίο εξετάσαμε είναι το τι έχουμε διαθέσιμο από τεχνολογικής πλευράς. Δηλαδή, Έχουμε το ABS ως σύστημα πέδησης χωρί εμπλοκή. Το σύστημα αυτό θεωρείται ότι είναι το πιο προηγμένο όσον αφορά τα συστήματα πέδησης. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες τεχνικές λύσεις που θα μπορούσαν να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα με μειωμένο κόστος για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Το άλλο ζήτημα για το οποίο θα ήθελα να πω κάποια πράγματα ακόμα είναι η περιβαλλοντική πτυχή και για το ζήτημα αυτό έχουμε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Σε αντίθεση όμως με άλλα οχήματα, όπως για παράδειγμα τα φορτηγά ή τα αυτοκίνητα, στην περίπτωση αυτή επικεντρωνόμαστε και πάλι στο ζήτημα των μοτοσυκλετών μετά από μια απουσία, αν θέλετε, νομοθετική στον τομέα αυτό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είχαμε επικεντρωθεί τόσο πολύ στον τομέα αυτό. Η νομοθεσία διαθέσιμη που έχουμε χρονολογείται από μία περίοδο αρκετά μακρινή και πιστεύω ότι θα πρέπει και εδώ, όπως έχουμε κάνει στα οχήματα, τα υπόλοιπα, να έχουμε μία ανάλογη νομοθετική πρωτοβουλία. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να πω είναι αυτό που είπατε και εσείς πριν από λίγο κύριε Πρόεδρε, ότι ε, υπάρχουν ε, πολλά διαφορετικά ζητήματα τα οποία εμφανίζονται όσον αφορά την ασφάλεια και την εξετάζουμε διαφορετικές κατηγορίες ε, οχημάτων. Η ασφάλεια δεν έχει να κάνει μόνο με τεχνικές απαιτήσει και προδιαγραφές. Έχουμε έρθει σε επαφή και με άλλες υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως για παράδειγμα τις αρμόδιες για την, για την κυκλοφορία με συγχωρείτε, ή τις υπηρεσίες αυτές που έχουν να κάνουν με το τεχνικό έλεγχο και τις άδειες Και το κάναμε αυτό προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή πρόταση που θα λαμβάνει υπόψη τις όλες τις επιμέρους απαιτήσει και που θα είναι ε, σε θέση να οδηγήσει σε ένα καλύτερο επίπεδο ασφάλειας και σε μια καλύτερη συνεκτικότητα ανάμεσα στα νομοθετήματα που ήδη υπάρχουν. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τους τεχνικούς ελέγχους, το ζήτημα αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο προς εξέταση στην πρότασή μας, αλλά έχουμε κάνει σχετικές ε, προτάσεις στο παρελθόν προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι ε, τα οχήματα θα έχουν τις τεχνικές εκείνες προδιαγραφές που θα επιτρέπουν μια πιο εύκολη και ομαλή έγκριση τύπου και που θα διευκολύνουν ουσιαστικά και όλη τη διαδικασία της εποπτείας. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να σας πω ότι ε, προσπαθήσαμε σε κάθε περίπτωση να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή ισορροπία και συνεκτικότητα με άλλες πρωτοβουλίες και άλλα νομοθετήματα τα οποία έχουμε γκρίνει στο παρελθόν που εξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαρτίνη. Σας ευχαριστούμε για την ε, βοήθειά σας και που αναφερθήκατε και στο ζήτημα του τεχνικού ελέγχου. Κύριε Κάμπα, κύριε Σιγητά, θέλετε να πάρετε τώρα το λόγο, θέλετε να κάνετε κάποιες τελικές παρατηρήσεις, θέλετε να αναφερθείτε επίσης στο χρονοδιάγραμμα και σε επισκέψεις που θα γίνουν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω του για τη συγκεκριμένη συνεισφορά. Στο έγγραφο εργασία που θα συζητήσουμε στι 28 Φεβρουαρίου, ήδη θα υπάρχουν περισσότερε λεπτομέρειε, θα είναι πιο πλήρη το έγγραφο. Θα ήθελα να κάνω κάποια ακόμη σχόλια. Καταρχήν σε σχέση με την ασφάλεια. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. τεχνικά μέτρα πράγματι μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια, όμως ε, η ίδια η συμπεριφορά ε, του, των ανθρώπων που οδηγούν ε, τις μοτοσυκλέτες είναι επίσης πολύ σημαντικό. Στις 8 Φεβρουαρίου το απόγευμα θα έχουμε ένα σεμινάριο για την ασφάλεια ε, των κινητήρων και τα τεχνικά μέτρα και ελπίζω οι σκιώδεις εισηγητές να μπορέσουν να συμμετάσχουν. Κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά στα συστήματα πέδησης, θα πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Είναι πολύ πλοκό. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια ισορροπημένη διατύπωση στο κείμενο. Όπως είπε και ο συνάδελφος από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς εγκαθιστούμε σε κάθε τύπο οχήματος. Ό,τι αφορά τις ε, μικρές σειρές, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά για μια ακόμη φορά να σας πω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε την καινοτομία στον τομέα των μοτοσυκλετών. Επίσης, ε, συνάδελφος αναφέρθηκε και στο εξωτερικό κόστος. Ε, είναι πολύ μεγάλο θέμα και αυτό για μας τις κατοχώρες. Εγώ ίσως να μην ασχολούμαι απευθεία με το θέμα του περιβάλλοντος, αλλά ε, ε, κοιτάξτε, εγώ έχω μοτοσικλέτα, έτσι λοιπόν ε, μπορώ να πω ότι ακόμη και ως χόμπι αν έχει κανείς μια μοτοσικλέτα και πάλι ρηπαίνει. Έτσι λοιπόν ε, οι ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες είναι μια πολύ μεγάλη υπόσχεση για το μέλλον ε, των πόλεων. Αν δούμε τι προβλήματα κυκλοφορίας έχουμε στις πόλεις, ε, αν έχουμε τέτοια μικρά μηχανάκια, ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, η ηλεκτρικά ποδήλατα, αυτή είναι μια δυνατότητα που δεν την έχουμε σκεφτεί ακόμη, πρέπει να τη συζητήσουμε εις βάθος. Την Παρασκευή, όχι την Πέμπτη κύριε Πρόεδρε, είναι η επίσκεψη μελέτης. Έτσι λοιπόν προσοχή, ε, να μην πάτε μια μέρα πριν την, την Παρασκευή είναι η σωστή ημέρα. Κατόπιν ε, είχαμε το σχόλιο από την κυρία Ρόιτοβα. σε επαφή από τους συναδέλφους από την Επιτροπή Τραν. Έχουμε τον συνάδελφο που είναι εισηγητής για την οδική ασφάλεια και εκεί αναφέρεται και το θέμα της πιστοποίησης. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά και να προσπαθήσουμε να έχουμε και μια καθολική προσέγγιση. Η πιστοποίηση και η ασφάλεια πρέπει να συμβαδίζουν, πρέπει να προχωρούν παράλληλα. Αυτά ήθελα να πω στη δεύτερη παρέμβασή μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. πολύ κύριε Φαντεκάμπ. Ε, να επιβεβαιώσω στα μέλη της Επιτροπής ότι το σχέδιό σας είναι. Θα δούμε το έγγραφο εργασία σας που αποτελέσει η βάση για τη συζήτηση που νομίζω θα παρουσιαστεί στις 28 Φεβρουαρίου, σωστά? Έχουμε κατόπιν ε, το σχέδιο έκθεση που θα πάει για μετάφραση 26 Μαρτίου. Θα συζητηθεί 14 ε, και 15 Απριλίου. 14 Μαΐου προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ε, ε, και τον Ιούνιο στην Ολομέλεια. Ε, θα συζητήσετε με παραγωγούς, με κατασκευαστές αυτοκινήτων, θα οργανώσετε μία εκδήλωση στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν ε, η βουλευτής, ε, οποιοδήποτε λοιπόν ενδιαφέρεται, είναι ευπρόσδεκτος. Επίσης, ε, έχουμε γνωμοδοτήσεις από την Επιτροπή Μεταφορών και την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η Επιτροπή Μεταφορών πιθανότατα να αναφέρεται στα θέματα που, σε αυτό που ανέφερε η κυρία ρότα σχετικά με τους ελέγχους των αυτοκινήτων ε, και επίσης ε, αν θέλει να συμμετάσχει κανείς στις ε, επισκέψεις που έχουν προγραμματιστεί είναι ε, Πιστεύω ότι θα τους προσκαλέσετε. Σας ευχαριστώ πολύ για το θέμα αυτό. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της καλής συνεργασίας. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μαρτινό από την Επιτροπή. Προχωράμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η έκθεση της κυρίας Κέπχαρτ σχετικά με την εφαρμογή της ε, οδηγίες για τις υπηρεσίε Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Είχαμε μια σειρά τροπολογιών ε, και συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών ε, και συζητήσεις για συμβιβασμούς. Θα δώσω τον λόγο στην κυρία Κέπχαρτ και να καλέσω και την κυρία Μαρία Μαρτιν Πράτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Θα της δώσω το λόγο για να συμμετάσχει και εκείνη στη συζήτησή μας η κυρία Χάνσλεκ είναι παρούσα, Λούκε Κάρτ, ο κύριο Κάμφερ δεν είναι παρόν. Εγώ είμαι παρόν, η κυρία Σουένσον και ο κύριος Σαλίνη δεν είναι παρόντες. Έχουμε αρκετούς κοιοδησίτες εδώ, αλλά δεν είναι όλοι παρόντες. Θα δώσω λοιπόν, πρώτα το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Εύελεν Κέπχαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους. Η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες ε, ε, έχει εμπνεύσει κάποιους από τους συναδέλφους μου. Αυτό είναι καλό. Και σε μια τόσο τεχνική έκθεση έχουμε λάβει τροπολογίες, κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα διότι δείχνει ότι το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδεις εισηγητές ε, για την ε, πραγματικά καλή συνεργασία. Είχαμε κάποιες διαφορές απόψεων, αυτό είναι ε, ε, απόλυτα φυσιολογικό από ε, πολιτικής πλευράς. Καταφέραμε όμως σε κάποια θέματα να διατυπώσουμε συμβαστικές τροπολογίες οι οποίες είναι σημαντικές. Θα ξεκινήσω με τους τρεις συμβιβασμούς μας, τις τρεις συμβαστικές τροπολογίες. Το ένα θέμα αφορά τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτηση στο σημείο 11 όπου μιλάμε για την προσβασιμότητα των κέντρων ενιαίως εξυπηρέτησης ε, δεν ε, υπήρχαν διαστάσεις απόψεων ως προς το περιεχόμενο. Είχαμε όμως τόσες ε, διαφορετικές προτάσεις. Πιστεύω ότι έχουμε βρει πολύ καλή διατύπωση ε, κατόπιν ε, προτάσεων του ΕΛΚ και των ε, φιλελευθέρων κάνουμε κάποιες προτάσεις σχετικά με τις μελλοντικέ εργασίες. όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα κέντρια ενιαίας εξυπηρέτησης που δεν προβλέπονται στην οδηγία περί υπηρεσιών είναι φυσικό όμω ότι τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν περισσότερε πληροφορίε από αυτέ που προβλέπονται στην οδηγία περί υπηρεσιών. Και εδώ μα ενδιαφέρει κυρίω η πληροφόρηση όσον αφορά το δίκαιο εργασίας Ε, τα οικονομικά θέματα, τον ΦΠΑ και άλλα σημαντικά και δεν μπορούμε να περιμένουμε ε, οι παροχοί υπηρεσιών να γνωρίζουν το δίκαιο των, κράτων, των κρατών μελών ε, σε αυτά τα θέματα. Είναι λοιπόν χρήσιμο να γίνεται κάτι τέτοιο. Και είπαμε ότι θα πρέπει να προβλέπεται βελτίωση όσον αφορά τις εργασίες των κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης σε πολλά κράτη-μέλη. Έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει ανάγκη βελτίωσης Κάνουμε λοιπόν έκκληση τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτηση να μην είναι μόνο μία ε, ψηφιακή πύλη. Θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι πίσω από αυτήν την πύλη οι οποίοι να παρέχουν πληροφορίες, ε, αλλά όχι μόνο να παρέχουν πληροφορίες, αλλά να μπορούν να βοηθήσουν και όσον αφορά τις εγγραφείοκρατικές διαδικασίες που πρέπει να ε, γίνουν. Είναι λοιπόν σημαντικό τα κέντρα εξυπηρέτησης πράγματι να εξυπηρετούν. Επίσης ε, σημαντικό είναι το θέμα της γλώσσας. Είχαμε μια μικρή συζήτηση μεταξύ μας ε, σχετικά με το ποια, ε, γλώσσα θα, σε ποια γλώσσα θα πρέπει ε, να γίνεται εξυπηρέτηση. Το πιο ωραίο θα ήταν σε 27 γλώσσες να γίνεται εξυπηρέτηση, αλλά αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το ζητήσουμε, Αυτό θα ήταν υπερβολικό για τις διοικήσεις των κρατών μελών. Ωστόσο, χρήσιμο θα είναι να γίνεται εξυπηρέτηση σε γλώσσες γενικά κατανοητές. Ε, τώρα τα φιλανδικά ή τα ελληνικά δεν είναι ε, συνηθισμένη η τα ελληνικα δεν ειναι συνηθισμενη γλωσσα στο, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αγγλικά και τα γαλλικά είναι πιο συνηθισμένες πιο, γλώσσες που χρησιμοποιούνται ευρύτερα. προτείνουμε στα κράτη-μέλη να ε, παρέχουν ε, ε, τις υπηρεσίες τους και στην γλώσσα της γειτονικής χώρας. Στο ΚΕΛ, για παράδειγμα, να υπάρχει εξυπηρέτηση και στα γαλλικά. Αυτά είναι που προβλέπονται στην ε, συμβαστική τροπολογία για το σημείο 11. Όσον αφορά το σημείο 12, εδώ διαπιστώσαμε και το, μας το είπαν ε, πολλοί από αυτούς που εργάζονται στα κέντρα ενίας εξυπηρέτησης. Είπαν ότι, ε, έχουν, ότι λαμβάνουν πολλά αιτήματα. Ναι, είναι ένα νέο μέσο Συγγνώμη, ότι δεν, έχουν, δεν λαμβάνουν πολλά αιτήματα. Πολλοί υπάροχοι υπηρεσιών δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν αυτά τα κέντρα ενιαία εξυπηρέτηση και γι' αυτό ε, καλούμε τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει εκστρατεία ενημερωτική ώστε οι υπάροχοι υπηρεσιών να ενημερωθούν ότι παρέχεται αυτή η δυνατότητα μπορούν να στραφούν στα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης και να λάβουν ε, πληροφορίες ε, σημαντικές. Πιστεύω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά θέματα στην έκθεση αυτή. Σημαντικό είναι δηλαδή τα μέσα που δίνουμε στους ε, παρόχους υπηρεσιών να ε, χρησιμοποιούνται σωστά, να μπορούν οι υπάρχοι υπηρεσιών να, λάβουν, να λαμβάνουν τι σωστές πληροφορίες ώστε να μην ε, ε, παίρνουν λάθος αποφάσεις όταν βρίσκονται σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Ε, μιλάμε για απλοποίηση της νομοθεσίας των κρατών μελών. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο σημείο που μα ενδιαφέρει στον τομέα αυτών. Η τρίτη συμβαστική τροπολογία ήταν αυτή που ήταν πιο δύσκολο να επιτευχθεί ε, φαίνεται στην τροπολογία η διαφωνία ε, των ε, πολιτικών ομάδων. Το θέμα εδώ ήταν η... το πεδίο εφαρμογής. Έπρεπε να δούμε αν υπάρχουν δυσκολίες ως προς τον ορισμό ή όχι. Καταλήξαμε όμως και εδώ σε μια πολύ σωστή ρύθμιση. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων προς ε, την κυρία Χάνσλικ και τον κύριο Λουκεγκάρτ ε, για την καλή συνεργασία. Και οι τρεις ε, κάναμε κάποιες υποχωρήσεις. Καταλήξαμε τελικά σε έναν πολύ καλό συμβιβασμό. Η κυρία Χάνσλικ είπε ότι η... Μπορώ να πω στην κυρία Χάνσλικ ότι μπορώ να δεχτώ και την τελευταία της τροπολογία σε, κάποια κράτη-μέλη, όχι σε όλα, γίνεται συζήτηση σχετικά με τον ορισμό της εξαίρεσης ε, των παρόχων υπηρεσιών. Και εδώ είχαμε τις ε, πιο σημαντικές δυσκολίες, αλλά η διατύπωση στην οποία καταλήξαμε το λαμβάνει αυτό υπόψη και πιστεύω ότι καταλήξαμε σε πολύ καλή διατύπωση και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που καταλήξαμε σε αυτή τη λύση. Στην αρχή πίστευα ότι δεν θα καταλήγαμε σε συμβιβασμό και ότι θα έπρεπε να ψηφίσουμε ε, και αυτό δεν θα ήταν πρόβλημα, αλλά καλύτερο είναι όταν δεν υπάρχουν διαφωνίες. Όσον αφορά τις τροπολογίες τώρα. Ε, έχουμε πολλές τροπολογίες, δεν θα αναφερθώ σε όλες, ε, διότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με πολλές από αυτές, δεν υπάρχουν προβλήματα. Μόνο για κάποιες πρέπει να πω ότι δεν συμφωνώ και θέλω να σας πω γιατί η πρώτη τροπολογία με την οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω είναι η τροπολογία του κυρίου Κομφέ, αριθμός 13, διότι η τροποποίησή του, κατά τη γνώμη μου, ε, βρίσκεται σε λάθος σημείο. Δεν αναφέρεται κατά τη γνώμη μου στο θέμα της ε, αξιολόγησης ε, αλλά στην διοικητική συνεργασία και θα ήθελα η τροποποίηση αυτή να μεταφερθεί στο σωστό σημείο. Το η δεύτερη τροπολογία στην οποία έχω πρόβλημα είναι η τροπολογία 22 του κυρίου Καράς. Δεν μπορώ να συμφωνήσω. Αύριο στην ε, συνάντηση των ε, συντονιστών θα συμφωνήσουμε να ανατεθεί η μελέτη σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης. Δεν νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο να προδικάσουμε τα αποτελέσματά της και να πούμε ότι η συστηματική αξιολόγηση είναι απολύτως θετική διότι αυτό δεν το θέλαμε τότε ως κοινοβούλιο. Συμπεριλήφθηκε επειδή ε, τα κράτη-μέλη ήθελαν οπωσδήποτε να συμπεριληφθεί. Είχαμε πει τότε ότι υπάρχει διαφωνία, θα το εξετάσουμε πιο προσεκτικά το θέμα. και θα εκφράσουμε θέση. Ε, εδώ ε, ταιριάζει και το θέμα των ε, πινάκων αντιστοιχία και αυτό έχει συζητηθεί έντονα στο Κοινοβούλιο. Δεν θα ήθελα λοιπόν να συμπεριληφθεί αυτό εδώ, όχι επειδή διαφωνώ, αλλά επειδή θα πρέπει να εξετάσουμε αν πράγματι είναι θετικό, θετική η συστηματική αξιολόγηση. Την τροπολογία 31 του κ. Λούκεγκάρντ επίσης δεν μπορώ να υιοθετήσω. Κύριε Λούκεγκάρντ. Ε, θέλετε ε, για το άρθρο 20 παράγραφος 2 ε, κατευθυντήρες γραμμές. Να σας θυμίσω ότι ως Κοινοβούλιο πετύχαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην μπορεί να υιοθετήσει κατευθυντήρες γραμμές σχετικά με την οδηγία αυτή. Αυτός ήταν ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εξέδωσε κατευθυντήρες γραμμές, αλλά εγχειρίδιο το οποίο δεν είναι νομικά δεσμευτικό. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να ζητάμε τώρα από την Κομισιόν κατευθυντήριες γραμμές τη στιγμή που στην ίδια την οδηγία ε, έχουμε ε, εμποδίσει κάτι τέτοιο. Αυτό θα ήταν ε, αντιφατικό από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάλκολμ, την τροπολογία σου υπαριθμών 38 δεν την έχω καταλάβει. Μήπως μπορείς να μου την εξηγήσεις. Εγώ είχα γράψει Ε, ότι θα πρέπει να συμμετέχουν οι, κοινωνικοί, οι κοινωνικοί εταίροι. Εσύ συμπεριλαμβάνει και τις επαγγελματικές Ε, Για μένα αυτοί, ε, ε, οι οργανώσει αυτέ συμπεριλαμβάνονται στους κοινωνικού εταίρους. Κοινωνικοί εταίροι για μένα είναι εργοδότες και εργαζόμενοι και γι' αυτό θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητη η προσθήκη αυτή. Αλλιώ θα πρέπει να απαριθμίσουμε όλου. αλλά θεωρώ ότι δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο ε, αν απλά αναφερόμαστε στους κοινωνικούς εταίρους. Δεν μπορώ να συμφωνήσω δεν ξέρω αν μπορείς να αποσύρεις ε, την ε, τροπολογία αυτή. Νομίζω ότι περιτεύει. Νομίζω ότι επρόκειται απλά για διευκρίνηση. Κοιτώ και τι υπόλοιπε τροπολογίε. Πραγματικά αναφέρομαι μόνο σε αυτέ ε, με τι οποίε έχω πρόβλημα. Με πολλέ από τι τροπολογίε δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μόρτεν. Ε, δεν μπορώ να συμφωνήσω και με την τροπολογία 69. Η ιδέα είναι καλή. Ίσως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάτι για την Ολομέλεια. Πρόβλημα έχω. Είμαι υπέρ της ηλεκτρονική ταυτοποίηση και εξακρίβωσης. Βρίσκω πολύ καλή την ιδέα αυτή, ωστόσο έχω πρόβλημα. Αν γράψουμε ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα δικά τους ηλεκτρονικά μέσα ταυτοποίησης εξακρίβωσης. Δεν ε, μπορώ να καταλάβω πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε κάτι τέτοιο. Όταν μιλάμε για ταυτοποίηση, εξακρίβωση της γνησιότητας, εάν στραφεί κάποιος ε, σε ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης ε, και χρησιμοποιεί δικά του μέσα, πώς το κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης μπορεί να γνωρίζει ότι δεν έχει γίνει εδώ κάποια ε, κατάχρηση ή παρατυπία. Ζητώ συγγνώμη, πολύ αργά το είδα αυτό, αλλιώς ε, θα το είχα αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα που συναντηθήκαμε. Αν ε, θέλεις να αποσύρεις την τροπολογία αυτή, μπορούμε να σκεφτούμε κάποια νέα διατύπωση για την Ολομέλεια, ώστε να μην έχουμε το πρόβλημα αυτό. Ε, αυτό έχω να πω, αλλιώς ε, θα πρέπει να καταψηφίσω την τροπολογία. Τροπολογία 70. Συμφωνώ με το πρώτο μέρος. Και εδώ θα ήταν χρήσιμο να διαγράψουμε το τελευταίο μέρος. Το όπως είναι η οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Ε, και εδώ πρόκειται για την λειτουργία του συστήματος ΙΜΗ, αλλά ε, ρητά αφαιρέσαμε από την οδηγία της υπηρεσίας την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Ε, η αναφορά αυτή θα οδηγήσει σε μια λανθασμένη πολιτική συζήτηση αν θέλουμε να συμπεριλάβουμε την οδηγία αυτή στο σύστημα ΙΜΗ. Αυτό θα πρέπει να γίνει μετά από συζήτηση για την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Ε, δείχνω, βρίσκω όμω ότι κάτι θα είναι προβληματικό. Μπορώ να δεχτώ λοιπόν την τροπολογία χωρί την ε, τελευταία αυτή προσθήκη. Αλλιώ θα την καταψηφίσω. Ε, θεωρώ ότι είναι προβληματική η τροπολογία αυτή, διότι αντίκειται σε αυτό που αποφασίσαμε στα πλαίσια τη οδηγία για τι υπηρεσίε. Να αποκλείσουμε δηλαδή από το πεδίο εφαρμογή στην οδηγία την απόσταση, απόσπαση εργαζομένων. Ε, κοιτάω τι σημειώσει μου. Νομίζω ότι αυτά είχα να πω. Α, υπάρχουν και κάποιες τροπολογίε του κυρίου Μούλτσερ, δεν είναι παρόν. Δεν θα αναφερθώ σε αυτές. Ε, είναι κάποιε που δεν μπορώ να δεχτώ, διότι Ε, ε, συνεπάγονται αποδυνάμωση της ε, οδηγίας για τις υπηρεσίες. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, θέλουμε θετική πολιτική για τους πολίτες. Θέλουμε κοινή αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό Ε, και όχι ε, να κοιτάμε τα εθνικά συμφέροντα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, γενικά μπορώ να δεχτώ ότι όλα τα υπόλοιπα, συμφωνώ με όλες τις άλλες τροπολογίες, αναφέρθηκα μόνο στα θέματα που θεωρώ προβληματικά για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε. Σας Σε ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γκέπχαρτ. Και όπως είπατε είναι πολύ θετικό το ότι τόσοι συνάδελφοι δείξαν ενδιαφέρον. Καταδεικνύει αυτό πόσο σημαντικό είναι να έχουμε εκθέσεις για, για την εφαρμογή οδηγιών στη δική μας την Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό το ότι καταφέρουμε να, καταφέρνουμε να δείξουμε αυτή τη στιγμή ότι όντως υπάρχει μια οδηγία και η εφαρμογή της οποίας θα πρέπει να είναι θετική βέβαια θα δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές. Στη συνέχεια θα απαντήσω και εγώ στα ερωτήματα τα οποία θέσατε. Και βέβαια οποιοδήποτε άλλος θέλει να πάρει το λόγο, η κυρία Βάιλερ ή οποιοδήποτε άλλος από την Επιτροπή, μπορούν να εγγραφούν στον κατάλογο ομιλητών. Η κυρία Χάνσλικ έχει πρώτη το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα Guardian ευχαριστήσω την Evelyn Gebhardt και όλους τους σκιώδεις ηγητές για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Σας ευχαριστώ για την διαλλακτική στάση που κρατήσατε, για το ότι θελήσατε να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες. Συμφωνούμε όλοι ότι η οδηγία αυτή είναι μία από τις πιο σημαντικές οδηγίες, είναι από τα πιο σημαντικά νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των παρόχων υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Χαίρομαι λοιπόν πολύ που βλέπω πώς βαίνει η εφαρμογή της οδηγίας αυτής σε όλα τα κράτη-μέλη. Σε ορισμένε χώρες, στο Λουξεμβούργο ε, και σε κάποιες άλλες, για κάποιους πολιτικούς λόγους, δεν καταφέραμε να δούμε την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Ωστόσο, τα περισσότερα κράτη-μέλη εφαρμόζουν την οδηγία αυτή Πράγμα το οποίο σημαίνει, αφού είπα και στην αρχή άλλωστε, ότι η οδηγία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για τι εταιρείε, για του παρόχου υπηρεσιών, για την ομαλή λειτουργία τη εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με όλε τι συμβαστικέ τροπολογίε που πρότεινε η Εύελιν. Όντω για το άρθρο 18 έγινε μια έντονη συζήτηση από ό,τι φαίνεται δεν καταλήγουμε εδώ πέρα σε κάποια, δεν καταλήγαμε σε κάποια συμφωνία. Ωστόσο θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εύελιν που δείχνει μια ανοιχτή διαλλακτική στάση για τη δική μας τη στάση και που αυτή τη στιγμή δέχεται να κοιτάξει και την δική μας την προσέγγιση για το άρθρο αυτό. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν την Εύελιν. Ε, οι συμβαστικέ τροπολογίε είναι πολύ καλέ και νομίζω ότι όλε οι πολιτικέ ομάδε θα είναι σε θέση να τι υποστηρίξουν. Όσον αφορά τα κέντρα νιές εξυπηρέτησης, συμφωνώ η ίδια προσωπικά και η δική μου πολιτική ομάδα απόλυτα με την πρόταση που έχει γίνει στο σημείο αυτό. Θεωρώ ότι τα κέντρα ενιαία εξυπηρέτηση είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα τη οδηγία. Έχουν συσταθεί, λειτουργούν. Το σημαντικό που θα πρέπει βέβαια να δούμε εδώ είναι ότι υπάρχουν κάποια περιθώρια βελτίωση στη λειτουργία του ορισμένα κράτη-μέλη. Και κάτι ακόμα. Όλε οι πληροφορίε που έχουν να κάνουν ε, με εκστρατείες προώθησης προϊόντων στα κράτη-μέλη, είναι πολύ σημαντικό να αξιολογούνται και από άλλα κράτη-μέλη. Είναι πολύ σημαντικό και στα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης να μπορούμε να έχουμε πληροφορίες που έρχονται από άλλα κράτη-μέλη. Είναι πολύ σημαντικό ένας πολίτης ο οποίος απευθύνεται στο κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης οποιαδήποτε, οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι σε θέση να έχει πρόσβαση και σε πληροφορίες που προέρχονται από άλλες χώρες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όλοι οι πολίτες, όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών να γνωρίζουν ότι έχουν πρόσβαση ισότιμη στα κέντρα αυτά ενιαίας εξυπηρέτησης. Το γλωσσικό το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό όπως καταλαβαίνετε σε οποιαδήποτε διασυνοριακή συνεργασία. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό στα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης να μην έχουμε μόνο τη γλώσσα της χώρας αλλά και των γειτονικών χωρών. Συνοψίζοντας υποστηρίζω με μεγάλη ευχαρίστηση τις συμβαστικές τροπολογίες της ε, εισηγήτριας και ως σκιώδη εισηγήτρια και εξ ονόματος πολιτικής μου ομάδας θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Εύελιν και τους υπόλοιπους σκιώδη εισηγητές. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή θα συμβάλλει σε μια καλύτερη εφαρμογή και λειτουργία της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Μια οδηγία που όπως σας είπα είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ουσιαστικά αν θέλετε το δικό μας το δημιούργημα γιατί η Επιτροπή ΙΜΚΟ είναι αυτή η οποία επεξεργάστηκε αυτή την οδηγία. Σα ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. ευχαριστώ και πάλι Εύελιν. Σας ευχαριστούμε και εμείς για την πολύ θετική αυτή ανταπόκριση. Κύριε Λέχαρτ, νομίζω ότι σας τέτησαν κάποιες ερωτήσεις. Όντως, καταρχάς να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με την εισηγήτρια και τους και οδησηγητές. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για, την, για το πολύ καλό αυτό σχέδιο έκθεσης και όπως είπατε και η ίδια, η όλη η εμπειρία, το όλο εγχείρημα ήταν πολύ θετικό και χάρηκα πάρα πολύ που είδα ότι καταφέραμε κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων να συμφωνήσουμε για ζητήματα τα οποία ήταν ιδιαίτερα επίμαχα από πολιτικής πλευράς. Ωστόσο πιστεύω ότι θα πρέπει να περάσουμε και στα επιμέρους σημεία τώρα, στις παρατηρήσεις που κάνετε για τις συγκεκριμένες τροπολογίες ξεκινώντας με την τροπολογία 31. Νομίζω ότι αναφερθήκατε σε αυτήν, έτσι δεν είναι. θα μπορούσα να δεχθώ την ε, διαγραφή της πρότασης που έχει να κάνει με, την, ε, με τις τη γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2011. Νομίζω ότι δεν συμφωνούσατε με το σημείο αυτό, δεν κάνω λάθο. Καλεί την Επιτροπή να εκδώσει το 2011 κατευθύνε γραμμές. Μπορώ να δεχθώ τη διαγραφή του σημείου αυτού, αν αυτό βοηθά τελικά την έβρεση ενός ε, μιας συμβαστική διατύπωσης. Θα μπορούσα να δεχθώ αυτή τη διαγραφή. Ας ε, περάσουμε τώρα στην τροπολογία 69. Είπατε ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε εκ νέου εδώ πέρα την διατύπωση. Θα μπορούσαμε εδώ πέρα να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια αξιολόγηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Αυτό θα επέλυε, πιστεύω, το πρόβλημα. Θα μπορούσατε να δεχτείτε κάτι τέτοιο. Στην τροπολογία 70 νομίζω ότι αναφερθήκατε. Έτσι δεν είναι. Το πρώτο τμήμα της τελευταίας πρότασης για το IMI. Το πρώτο αυτό τμήμα στο οποίο λέγεται ότι ε, το IMI μπορεί να χρησιμοποιείται για άλλες σχετικές οδηγίες. Θα ήθελα να διατηρήσουμε το σημείο αυτό. Το τελευταίο τμήμα της πρότασης, δηλαδή όπως είναι η οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων, νομίζω ότι το σημείο αυτό μπορούμε να το διαγράψουμε. Νομίζω ότι αυτό αποτελούσε ένα συμβιβασμό και στην περίπτωση αυτή θα μπορούσα να δεχθώ και την πρότασή σας. Αυτά είχα να πω για τις επιμέρους ε, τροπολογίες. Δεν θα ήθελα να επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή για τις άλλες προτάσεις που έχουν γίνει. Υποστηρίζουμε όλες τις συμβαστικές τροπολογίες και ουσιαστικά την πλειοψηφία των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λακίγκαρτ, κάποια σχόλια και από μένα. Καταρχήν για την τροπολογία 38 να απαντήσω, την έχω συμπεριλάβει γιατί ξέρω ότι η πρακτική σκοπιά Ήδη υπάρχουν πάρα πολλέ επικοινωνικέ ενώσει σε περιφερειακό επίπεδο, όπω τα εμπορικά μιλητήρια που ήδη εμπλέκονται σε ό,τι αφορά την παροχή πληροφοριών στις επιχειρήσεις ε, για την οδηγία για τις υπηρεσίες και πολλές φορές ε, παρέχουν ε, και πληροφορίες για τις συμβάσεις. Έτσι λοιπόν, απλώς ε, ήθελα να τονίσω εδώ ότι συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό και οι επαγγελματικές ενώσεις. Όμως συμφωνώ ότι όλοι οι οικονομικοί φορείς πρέπει να εμπλέκονται και κυρίως ε, σε χώρες όπου υπάρχουν ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης, κοινωνικής εταιρικής σχέσης. Έτσι λοιπόν, ε, ε, ίσως αυτή η τροπολογία να μην ε, είναι το κατάλληλο συμπείο να μπει εδώ. Δεν θα επιμείνω. Τώρα, αν μπορώ να βοηθήσω την, για την ερώτηση του κ. Λουκέγκαρτ, ξέρουμε ότι η Κομισιόν αναθεωρεί την οδηγία της ηλεκτρονικής υπογραφής για να υπάρχει ένα κοινό σύστημα ε, επαλήθευσης έτσι ώστε να δίνεται αδειοδότηση για την παροχή υπηρεσιών και νομίζω ότι υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα να έχουμε αμοιβαία αναγνώριση ε, των ηλεκτρονικών υπογραφών αν δεν έχουμε ήδη την πλατφόρμα σε σχέση με την ηλεκτρονική υπογραφή. Έτσι λοιπόν ε, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να προωθήσουμε αυτό το θέμα της πλατφόρμας καταρχήν και για το ίμι το σύστημα ΙΜΗ δίκιο έχετε να λέτε ότι δεν αφορά μόνο την οδηγία της υπηρεσίας. Έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ και στο θέμα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Έτσι λοιπόν, ίσως δεν χρειάζεται να αναφέρουμε την απόσπαση των εργαζομένων συγκεκριμένα, αλλά είναι αλήθεια ότι είναι ένα μηχανισμός που χρησιμοποιείται και εκτός της οδηγίας των υπηρεσιών. Όμως, ε, σας κάλεσε σε μια συνδιάσκεψη της Κομισιόν την Πέμπτη όπου θα συζητηθούν ε, οι επιπτώσεις ε, του συστήματος ΙΜΗ και η συνέπεια στο πλαίσιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Είναι ένας ε, σημαντικός μηχανισμός που χρήζει υποστήριξη. Και επίσης νομίζω ότι η υποστήριξη που δίνουμε, η πολιτική υποστήριξη που δίνουμε στα κράτη-μέλη, για να ε, υποστηρίξουν οικονομικά αυτό το μηχανισμό είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να το αναγράφουμε εδώ σαφώς. Και νομίζω ότι για το θέμα της αμοιβές αναγνώρισης και για το θέμα της αξιολόγησης ομοτήμων πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτό συμπεριλαμβάνεται η σχετική αναθεώρησή του και η εφαρμογή του σε άλλες πτυχές της οδηγίας για την ενιαία αγορά συμπεριλαμβάνονται στο Single Market Act. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή θα πρέπει να το διερευνήσουμε αν θα είναι στο ορθό πλαίσιο, τώρα αν εδώ είναι πρώιμο αυτό θα πρέπει να το δούμε. Κατά τα λοιπά νομίζω ότι η έκθεση μπορεί να είναι πολύ καλή και ευχαριστώ την εισηγήτρια που έχει δεκτεί ορισμένες από τις τροπολογίες γιατί έχουμε ιδιαίτερη προσθεμένη αξία εδώ. Κυρίες Βάιλα και Τάιλα, δίπλα κάθοντα σήμερα, καταρχήν κυρία Βάιλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα είναι πολύ καλά, καλό το ότι ε, το αναφέρατε κι εσείς. Ε, μου έκανε εντύπωση διότι παρακολούθησα τη συζήτηση από την αρχή. Όταν υιοθετήθηκε η οδηγία, ζητήσαμε ήδη τότε να υπάρξει μια ε, εντατική και εκτενής εκστρατεία πληροφορίας. Τώρα, από την πλευρά της Κομισιόν, τώρα το ξαναζητάμε. Τι έγινε τα τελευταία δύο χρόνια. Διαπιστώνω ότι ομάδες ενδιαφερόμενες όπως είναι τα επιμελητήρια, ε, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια ε, ή τα εμπορικά επιμελητήρια της ε, Γερμανίας δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση. Οι κυβερνήσει όμως που επίσης θα έπρεπε να έχουν ασχοληθεί με το θέμα δεν έχουν κάνει ούτε αυτές ε, καμία εκστρατεία για ένα τόσο σημαντικό πολιτικά θέμα. Όταν σκέφτομαι το τι έγινε πριν ε, δύο-τρία χρόνια στην ε, Γαλλία, στη Γερμανία, θεωρώ ότι θα, θα είχε φανεί χρήσιμο εάν είχε γίνει μια γενική εκστρατεία σχετικά με τις συνέπειες, το νόημα, ε, τα προβλήματα της ενιαίας αγοράς. Η Κομισιόν θα έπρεπε να κάνει μια τέτοια εκστρατεία και όχι να το αφήσει αυτό στα κράτη-μέλη. Πράγμα που συνέβη τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Ε, στην Πολωνία ακούω έχουν γίνει πολλά. Στην Γερμανία διαπιστώνω ότι οι διάφορε ενώσει ε, που καταρτίζουν οι ίδιες τα μέλη του έχουν κάνει κάτι, αλλά αυτό δεν αρκεί. Ναι, νομίζω ότι με επεκτεύεται για το ότι τα κρατημέλη δεν ε, έχουν προωθήσει αυτό το θέμα ε, τόσο αυστηρά όπως σημείωσα και εγώ στην κυβέρνηση μου χθες κύριε Τάιλεν ευχαριστώ, ευχαριστώ και την Ευελίν για όλη τη δουλειά της και ευχαριστώ και τους προηγούμενους ομιλητές για τα σχόλια Λοιπόν, σε σχέση με όσο είπε η Μπάρμπαρα, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα Είναι καλό όταν ψηφίζουμε νομοθεσία να την αναφερούμε και να βλέπουμε την εφαρμογή της για τα κέντρα ενέας εξυπηρέτησης ε, πρέπει να δούμε γιατί σε ορισμένα σημεία λειτουργούν ενώ σε άλλα μέρη όχι. Ο Μάλκον ανέφερε κάτι και για τους σπόρους. Ε, όταν περάσαμε την νομοθεσία του 2006 δεν μπορούσε, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την παγκόσμια κρίση. Πρόκειται εδώ για μια νομοθεσία που αφορά το 70% του ΑΕΠ, τις υπηρεσίες στο μέλλον, θα είναι έτοιμο μηχανή της ανάπτυξης και αναφερθήκατε, Μάλκομ, ε, στους πόρους τα κρατεμέλη. Ξέρουμε ότι πολλά κρατεμέλη προβαίνουν σε περίπεκοκές, έτσι λοιπόν αυτό έχει και αντίκτυπο ε, στα κέντρα ενέσης εξυπηρέτησης. Νομίζω ότι καλό θα ήταν εμείς να πιέσουμε τα κράτη-μέλη για να εκταμιεύσουν αυτούς τους πόρους, ε, γιατί έτσι θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν τα επιχειρηματικά μοντέλα, να δημιουργήσουν δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να αναπτυχθούν οικονομίες. Και τώρα για τη συνάντηση της Πέμπτη, καλό θα ήταν να έχουμε κάποιο feedback σχετικά με το πώς λειτουργεί το ΙΜΗ. Η Εύελιν το ανέφερε στο επεξηγηματικό σημείο με αυτό. Νομίζω ότι είναι σημαντικό πράγματι να έχουμε feedback ως Επιτροπή για το τι συμβαίνει, γιατί αν είμαστε σοβαροί και μιλήσαμε για ηλεκτρονικές υπογραφές και και εδώ ε, έρχεται και το ψηφιακό θεματολόγιο. Αν δεν έχουμε ψηφιακοποίηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώ θα λειτουργήσουν στην πράξη οι ηλεκτρονικέ επιγραφέ και πώ θα γίνουν όλε αυτέ οι διασυνδέσει. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι είναι σημαντικό να το συζητήσουμε αυτό στην Επιτροπή, να προωθήσουμε τη στρατηγική μα, να δώσουμε στι υπηρεσίε ε, την προτεραιότητα που του αρμόζει. Και πραγματικά ε, νομίζω ότι η όθηση που δίνουμε σε αυτή την Επιτροπή είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να λειτουργούν ορθά υπηρεσίε και να αποτελούν μηχανή για την δημιουργία θέσεων εργασία. Ευχαριστώ κύριε Τάιλερ. Η διάσκεψη τη Πέμπτη θα απαντήσει κάποιε από τι ερωτήσει σα για το email. Ίσως για κάποια τελευταία σχόλια να δώσω το λόγο στην κυρία Μάρτιν Πράτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό από τη δική μας πλευρά είναι να ευχαριστήσουμε το Κοινοβούλιο για την εξαιρετική δουλειά του και να τονίσουμε πόσο χρήσιμε είναι τέτοιε εκθέσει. Στο παρελθόν, πολύ συχνά, μετά από τι διαπραγματεύσει, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, ξέχασαν τι, ξεχνούν τι συμβαίνει στην πράξη με τι οδηγίε, όμω ε, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε πλέον, ε, γιατί χάνουμε την αξιοπιστία μα ε, και δεν ξέρουμε πολλέ φορέ τι συμβαίνει με κάποιε οδηγίε τρία-τέσσερα χρόνια μετά την ψήφισή του. Έτσι λοιπόν, αυτό το έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα όταν μιλάμε για μια τέτοια νομοθεσία όπως η οδηγία για τις υπηρεσίες. Ορισμένες από τις προτάσεις ε, και κάποια από την πίεση που βάλετε στην έκθεση της κυρίας Κέμπαρτ ε, είναι πάρα πολύ χρήσιμες ε, και για τη δουλειά που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε με τα κράτη-μέλη. Αναφερθήκατε πολύ στα κέντρα ενιαία εξυπηρέτησης πράγματι. Μόνο με την άσκηση πίεση στα κράτη-μέλη, τα κέντρα ενιαία εξυπηρέτησης θα γίνουν αυτό που πρέπει να γίνουν, δηλαδή εθνικά ηλεκτρονικά κέντρα διακυβέρνηση για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις, για του αυτοπεσχολούμενου για τη διοίκηση, όλους αυτούς θα τους εξυπηρετήσουν ε, ε, με ένα πολύ πιο γρήγορο, λιγότερο γραφειοκρατικό τρόπο και μπορούν να έχουμε και διασυνοριακή χρήση. Έτσι λοιπόν πρέπει να εργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι αναγνωρίζονται οι ηλεκτρονικές επιγραφές και η ηλεκτρονική ταυτοποίηση αναγνωρίζεται όταν χρειάζεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, τμήμα των εργασιών μας που προωθείται και έχουμε μία σειρά διαδικασιών ε, για την ταυτοποίηση και για την επαλήθευση. Έτσι λοιπόν μην ξεχνάμε ότι και αυτή η δουλειά πρέπει να προωθεί με τα κράτη-μέλη και είναι σημαντική και για τα σημεία επικοινωνίας ε, η πίεση μπορούμε να ασκήσουμε στα κράτη-μέλη είναι ευπρόσδεκτη. Η Κομισιόν από τη δική της πλευρά έκανε όσα δύνατο και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από την παραγωγή Φιλανδίων και τη μετάφραση σε όλες τις επίσημες γλώσσες ε, μέχρι την παραγωγή βίντεο για να προωθήσουμε τα κεντρινές εξυπηρέτηση. Δημιουργούμε εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη. Ας μην ξεχνάμε το πιο αποτελεσματική επικοινωνία για τους χρήστες των κέντρων εξυπηρέτηση πρέπει να γίνει σε εθνικό, τοπικό, περιφερειακό επίπεδο. Έτσι λοιπόν ε, αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί από εμά. Πρέπει να γίνει από τα κράτη-μέλη αυτή η προσπάθεια. Και επίσης η δημοσιονομική κατάσταση πολλών κρατών είναι δύσκολη. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε να διαδίδουμε τις πληροφορίες για τα κέντρα εξυπηρέτηση, γιατί διαφορετικά θα, θα υπάρχει κανένα. Και ένα άλλο μέτωπο που ασκείται πίεση και εμεί καλωσορίζουμε είναι στο τομέα της διοικητικής συνεργασίας ε, για το IMI. Γιατί, γιατί αν δεν ε, υποστηρίξουμε τις προσπάθειες για την κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων και των χρηστών του IMI σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αυτό το εργαλείο συνεργασίας μεταξύ των δικήσεων, διαλόγου μεταξύ διάφορων κρατών μελών δεν θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τον έλεγχο της ασφάλειας και την ποιότητα των υπηρεσιών και τις διασυνοριακές υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν είναι πολύ χρήσιμο το μήνυμα που συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο έκθεση του Κοινοβουλίου. Σε αυτό το στάδιο η Κομισιόν ε, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ευχαριστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το επικοινωνικό έργο του. Ελπίζω να συνεχίσετε να μας βοηθείτε, να ασκήσουμε πίεση και να σημειώνουμε πρόοδο γιατί ακόμη δεν έχουμε ολοκληρώσει το έργο μα. Σα ευχαριστώ. Good. Um, Σας ευχαριστούμε. Εβελίν, θέλεις ε, να κλείσεις τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχήν, είναι σημαντικό σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παίρνουμε στα σοβαρά τη δουλειά μας. Με την οδηγία περί υπηρεσιών ε, έχουμε ιδιαίτερο τέτοιο χρέος διότι εμείς ε, βγάλαμε κάτι λογικό από την πρόταση της Κομισιόν το οποίο να λειτουργεί στην πράξη. Τη δική μας πρόταση υιοθέτησαν τελικά οι Υπουργοί στο Υπουργικό Συμβούλιο και γι' αυτό μας ενδιαφέρει να δούμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη με αυτό. Νομίζω ότι πρόκειται για υποχρέωσή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, για τις ε, παρεμβάσεις τους. Ε, θα συνεννοηθώ με τον Μόρτεν Λίκεκάρτ. Ίσως θα μπορέσουμε μέχρι αύριο να βρούμε κάποια λύση. Να ευχαριστήσω την Μπάρμπαρα για την έκκληση της σχετικά με την παροχή πληροφοριών. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό ότι τα κράτη-μέλη φαίνεται να μην ε, διατίθενται να ε, κάνουν μια εκτενή ε, εκστρατεία πληροφόρησης αλλά Είναι και ένα πρόβλημα το ότι δεν εγκρίνατε τότε την ιδέα μου να υπάρχει συντονισμός των διαφόρων ε, ε, εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, το ΕΛΚ τότε είχε αντιτεθεί στην ιδέα αυτή. Έπρεπε λοιπόν να την απεμπολίσουμε. Νομίζω όμως ότι όλοι σήμερα βλέπουμε ότι δεν ήταν καθόλου κακή η ιδέα. Βρίσκω ότι είναι κρίμα ότι δεν με ακολουθήσατε τότε στο θέμα αυτό. Ήταν όμως άλλα θέματα τότε πιο σημαντικά, γι' αυτό και εγώ είχα παραιτηθεί από την ιδέα. Και όσον αφορά τα ε, Κάθριν, τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης, γιατί δεν έχουν... Ε, γιατί δεν λειτουργούν καλά. Αυτό είναι θέμα των κρατών μελών. Ε, Εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει τουλάχιστον να το ρωτήσουμε αυτό, να το ερευνήσουμε. Και ε, γι' αυτό ε, ε, ε, αυτό το θέμα είναι το μεγαλύτερο μέρος της εκθεσής μου και γι' αυτό υπάρχουν και περισσότερες τροπολογίες. Είναι ο πυρήνας της οδηγίας περί υπηρεσιών. θα πρέπει να ε, γίνεται σεβαστό το δίκαιο της χώρας ε, στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες αλλά θα πρέπει να παρέχονται και σωστές πληροφορίες προς τους παρόχους υπηρεσιών ε, για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό ήταν η σημαντική τροποποίηση του άρθρου 16. Ήταν σημαντικό λοιπόν να δημιουργηθούν τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης για να υπάρχει καλή ισορροπία. Μάρκολμ, ήδη έχω μακρηγορήσει, ζητώ συγγνώμη αλλά όταν αρχίζω να μιλάω για την οδηγία περί υπηρεσιών ε, δεν σταματάω. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι και εμείς ε, συμμεριζόμαστε τον ενθουσιασμό σου. Δεν ε, παραπονιέμαι λοιπόν και νομίζω ότι είναι χρήσιμο να βοηθήσουμε όσο μπορούν τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι και η κυρία Μάρτιν Πράτ νιώθει ότι οι προσπάθειες της, Επιτροπή, της Επιτροπής ενισχύουν το θέμα αυτό σε εποχή ε, μειωμένης ε, οικονομικής ανάπτυξης ε, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε προτεραιότητα στα θέματα που μπορούν να βοηθήσουν την κατάσταση. Θα δώσω στην κυρία Κόμη την έκθεση, τη δυνατότητα στην κυρία Κόμη την Προεδρία για τα επόμενα δύο θέματα. Ε, επόμενο θέμα είναι η έκθεση του κυρίου Καράς. θα της δώσω λοιπόν θα της αναθέσω την Προεδρία. Θα επανέλθω για να κλείσω την ε, πρωινή συνεδρίαση. Παρακαλώ.

Εγώ θέλω να ξεκινήσω το δεύτερο μέρος με την πράσινη βίβλο για την διακυβέρνηση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Εδώ έχουμε μία σειρά συνδικών γιατί υπήρξαν κάποιες τελευταίες στιγμής τροπολογίες και δεν ε, τις έχω διαθέσιμε σε όλες τις γλώσσες. Έτσι λοιπόν λείπουν οι μεταφράσεις, αλλά θα διαβαστούν σήμερα από τη γραμματεία την ώρα του γεύματος. Έτσι λοιπόν, κατόπιν αυτής της ε, υπηρεσιακής ανακοίνωσης, εγώ θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Κάρας για να μας ε, παρουσιάσει τη γνωμοδότησή του. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στην καρέκλα του Προέδρου. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ήδη υπόθηκε, ασχολούμαστε τώρα με μια γνωμοδότηση της Επιτροπής ΙΜΚΟ για την εταιρική διακυβέρνηση. Η αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή είναι η Επιτροπή ΕΚΟΝ. Προσπάθησα να να ενσωματώσω στην έκθεση της ΕΚΟΝ κάποιες τροπολογίες που έχουμε, ε, ώστε και από τις δύο πλευρές να ε, περάσω τις θέσεις μας. Ε, τώρα συζητάμε μια γνωμοδότηση και το βασικό της μήνυμα είναι ότι η οικονομική κρίτη έχει δείξει κάποιες ε, σημαντικές αδυναμίες ε, στην διακυβέρνηση των χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων. Η βασική ενδιαφερόμενη, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι αρχές εποπτείας θα πρέπει να κάνουν περισσότερα πράγματα. Θα πρέπει να έχουμε ε, συνέστηση της ε, ευθύνης απέναντι στους ε, μετόχους. Θα πρέπει να υπάρχουν συστήματα ελέγχου και αντιστάθμισης. Θέλω πρακτικές αλλά νομικά δεσμευτικές ρυθμίσεις στην γνωμοδότηση την οποία έχετε λάβει κάποια από εσά στη δική σας γλώσσα, άλλοι τις έχετε λάβει στα αγγλικά. Επικεντρωνόμαστε σε επτά σημεία. Καταρχήν ε, στο θέμα της αναλογικότητας ε, των ε, ρυθμίσεων. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο τύπος του χρωματοπιστωτικού ιδρύματος, εάν μιλάμε δηλαδή για ιδιωτική τράπεζα καταθέσεων ή για τράπεζα επενδύσεων, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος, η για τραπεζα επενδυσεων ωστε να λαμβάνετε υποψη το μεγεθος η λειτουργια και το μοντέλο της επιχείρησης. το διοικητικό ε, Συμβούλιο θα πρέπει να υπόκειται σε εποπτεία, θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός. Δεύτερον, το ε, Εποπτικό Συμβούλιο δεν θα πρέπει μόνο βραχή πρόθεσμα να λαμβάνει υπόψη το συμφέρον ε, των ε, καταθετών. Θα πρέπει και μακροπρόθεσμα να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα του Ιδρύματος. Τρίτον, χρειαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, ισχυρά μέτρα για την ε, πρόληψη των ε, συγκρούσεων συμφερόντων. Τι σημαίνει αυτό να μην υπάρχουν ασύμβατες δραστηριότητες για παράδειγμα συμβουλή σχετικά με τις επενδύσεις και ταυτόχρονα διαχείριση κάποιων ταμείων. Αυτά θα πρέπει να διαχωρίζονται. Ε, θα πρέπει να ρυθμίζονται ε, οι συγκρούσεις συμφερόντων και θα πρέπει να υπάρχουν ε, ενιαίοι κανόνες στην Ευρώπη. Το τέταρτο σημείο έχει να κάνει με το ότι τα ανώτερα στελέχη και το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να, να είναι νομικά υπόλογοι για τη σωστή υλοποίηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης όχι μόνο ε, τα ανώτερα στελέχη. Τα, ανώτερα στελέχη. Επίσης, όσον αφορά την διαχείριση κινδύνου, οι συμμετέχοντες ε, στο θέμα αυτό ε, δεν έχουν καταλάβει ποια είναι η ευθύνη τους. Θα πρέπει να Υπάρχουν ε, οι υποχρεωτικές επιτροπές κινδύνους, board risk committees. Θα πρέπει να δημιουργηθούν αυτές οι επιτροπές. Έκτον, οι θεσμικοί επενδυτές θα πρέπει να συμμετέχουν στον διάλογο με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να υπάρχουν ε, καλοί κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης ε, και να ε, διασφαλίζεται το συμφέρον των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι θεσμικοί επένδυτες θα πρέπει να τηρούν έναν διεθνή κώδικα ορθής πρακτικής. Το τελευταίο σημείο της νομοδότησής μου ε, είναι μια παραπομπή στο CRD3, την οδηγία για τις κεφαλαιακές ε, Εδώ έχουμε καθορίσει κανόνες ε, σχετικά με την πολιτική αποδοχών. Θέλουμε στα επενδυτικά κεφάλαια να υιοθετηθούν οι κανόνες αυτοί και όσον αφορά την καλή διακυβέρνηση θα πρέπει ε, να υπάρχει ε, παραπομπή στην οδηγία της κεφαλικής απαιτήσει και την ε, πολιτική αποδοχών. Αυτά είναι τα βασικά σημεία στην γνωμοδότησή μου. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Σήμερα Θα λάβουμε την πρόταση της νομοδότησης σε όλες τις γλώσσες, ε, θα τη συζητήσουμε και θα την ψηφίσουμε στις 28 Φεβρουαρίου. Σας ε, ευχαριστώ θερμά. Παρακαλώ να ακούσω τις παρατηρήσεις σας. Ε, παρακαλώ και να υποστηρίξετε την πρότασή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κάρας. Θα δώσω τώρα το λόγο στους κοιόδης συζητητές. Βάλε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Καράς. Ε, πριν 10 λεπτά έλαβα την γερμανική μετάφραση, αλλά δεν είναι τόσο πολύπλοκο το θέμα. Ε, ήδη είχα διαβάσει το αγγλικό κείμενο και κατάλαβα τι ζητάτε. Αυτά που μας είπατε τώρα εδώ προφορικά ε, με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνοι. Αλλά να πω ανοιχτά ότι δεν βλέπω αυτά που είπατε να αντικατοπτρίζονται στο κείμενό σας, διότι το κείμενό σας είναι πολύ θολό. Τα ρήματα, τονίζει, αναγνωρίζει, Εσείς μας είπατε ότι θέλετε κάτι νομικά δεσμευτικό και κάτι πρακτικό, πραγματοποιήσιμο. Αυτό δεν βλέπω να αντικατοπτρίζεται στο έγγραφό σας. αλλά εάν επιμείνετε σε κάτι ε, νομικά δεσμευτικό θα ε, σας υποβάλω σχετικές τροποποιήσεις. Ε, επίσης, σε όσον αφορά κάποια θέματα, μάλλον έχουμε καθυστερήσει από την Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων. Έχουμε την οδηγία για τα ίδια κεφάλαια. Ε, ε, τα κράτη-μέλη έχουν δικούς τους ε, κανόνες. Η Γερμανία ήδη έχει κάτι για τα εποπτικά συμβούλια. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει κάνει κάποια πράγματα σχετικά με τα μπόνους. Το ότι συζητάμε τώρα μια πράσινη βίβλο σημαίνει ότι έχουμε καθυστερήσει ήδη δύο χρόνια και μιλάμε για μία πράσινη βίβλο που λαμβάνει υπόψη τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Για την άλλη πλευρά θα ε, έχουμε άλλη νομοθεσία η οποία, είναι, η οποία φτάνει πολύ αργά. Ε, στο παρελθόν ε, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι είχαμε λάθος κίνητρα όχι μόνο όσον αφορά τα ανώτατα επίπεδα των μεγάλων επιχειρήσεων και όσον αφορά τον μεγάλο όγκο ε, ξέρουμε ότι έχουν πληρωθεί πολλά μπόνους ε, ε, σε σε εκτενέστερη ομάδα και στη Γερμανία και στην Αυστρία όσον αφορά τους καταναλωτές. Θα πρέπει να αναφερθεί αυτό και στην δική σας Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εσάς θα ήθελα να ακούσω περισσότερα διότι ε, έχουν επηρεαστεί αρνητικά οι καταναλωτές. Αυτές είναι οι βασικές μου παρατηρήσεις ε, όσον αφορά δηλαδή τα όσα είπατε, ε, εντάξει τα δέχομαι, αλλά την επιτροπή που θα, συγγνώμη την πρόταση που υποβάλλουμε στην Επιτροπή Οικονομικών θα πρέπει να την διατυπώσουμε πιο σαφώς. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλοι σκιώδεις εισηγητές στην αίθουσα, να ξεκινήσουμε με τη συζήτηση. Ντεγιόν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η γνωμοδότηση που έχει υποβάλει ο κύριος Κάρας αποτελεί καλή βάση. Συμφωνώ με τα όσα είπε η Μπάρμπαρα Βάιλερ ότι θα μπορούσε να ενδυναμωθεί σε κάποια τη σημεία, αλλά είμαι ικανοποιημένος με τον προσανατολισμό, με την κατεύθυνση που ακολουθεί η γνωμοδότηση αυτή Οι τροπολογίε μου θα έχουν να κάνουν με τέσσερα σημεία. Πρώτον, μια γενική παρατήρηση. Θεωρώ ότι η εισαγωγή είναι καλή, ωστόσο θα πρέπει να λέμε εδώ ότι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί επηρεάζουν επίσης και τους φορολογούμενους, γιατί οι φορολογούμενοι ουσιαστικά πρέπει να πληρώσουν για τους οργανισμούς αυτούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν το ζήτημα αποκτά και κοινωνικές διαστάσεις σημαντικές. Δεύτερον, δεν γίνεται καθόλου λόγος για τους εξωτερικούς ελεγκτές, ότι αυτοί αναφέρονται στην πράσινη βίβλο. Θεωρώ ότι και οι εξωτερικοί ελεγκτές και ο έλεγχος που κάνουν θα πρέπει να τονίζεται στο κείμενο. Τρίτον, δεν γίνεται πουθενά μνήα στο ρόλο των εργαζομένων. Γιατί και αυτοί με τη σειρά τους, οι υπάλληλοι δηλαδή, μπορούν να συμβάλλουν στα μακροπρόθεσμα συμφέροντα τα οποία θέλουμε εμείς να προασπίσουμε. Τέταρτον, συμφωνώ με αυτό που η κυρία Βάιλερ όσον αφορά τα μπόνους. Σαφώς υπάρχουν και άλλες Γίνεται εδώ πέρα μια αναφορά στο CRD3, στην οδηγία για τι κεφαλαϊκέ απαιτήσει. Το δέχομαι αυτό. Ωστόσο το ζήτημα των πόνου είναι πολύ σημαντικό. Στον Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ληφθεί κάποια μέτρα. Κάποια στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών είπε ότι δεν ήθελε να προχωρήσει πάρα πολύ με το μέτρο αυτό γιατί θα μπορούσε να συλλέξει, είπε, πάρα πολλά χρήματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν υπάρχει απαραίτητη βούληση για την αντιμετώπιση του ζητήματο αυτού που οδηγεί ουσιαστικά σε έντονη κοινωνική ένταση. Βλέπουμε ότι αυξάνεται από τη μια η φτώχεια και αυξάνονται από την άλλη και τα μπόνους. Νομίζω ότι και αυτό το ζήτημα θα πρέπει να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντιγιόνγκ Στάιλερ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον συγκεκριμένο Συμφωνώ με τους υπολείπους. Πιστεύω ότι είναι μια καλή αφετηρία για τις συζητήσεις μας και ευχαριστώ τον κύριο Κάρας. Αν δείτε τις επισημάσεις του, ορισμένα θέματα αλληλοσυνδέονται, κυρίως χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για καλή και ανάγκη για καλύτερη διακυβέρνηση των εταιριών. όμω, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί πριν ε, την κρίση είχαν ε, συστήσει εταιρικές ε, και εταιρική διακυβέρνηση και ήθελα να ρωτήσω γιατί αισθάνονται τόσο άσχημα για το θέμα αυτό. Ποια είναι τα κυρία ζητήματα. Εμείς έχουμε εργαστεί πολύ για την εταιρική ευθύνη σε αυτό το κοινοβουλίο για την κοινωνική εταιρική ευθύνη και μπορώ να πω ότι υπάρχουν διάφορες πολιτισμικές διαφορές αλλά έχουμε και την παράγραφο 3 για τους μετόχους και τους μεριδιούχους. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα κύρια σημεία. γιατί πρέπει να μιλήσουμε για τα συμφέροντα των μεριδιούχων ε, ή πρέπει να δούμε την ευρύτερη κοινότητα των μετόχων. Ε, και πρέπει να δούμε το θέμα της διακυβέρνησης. Ένα από το θέμα που πρέπει να συζητήσουμε είναι ε, το μακροπρόθεσμα συμφέροντα του Ιδρύματος, γιατί όπως είπε και η Μπάρμπαρα, αυτό συμφέρεται με το θέμα των αποδοχών και των πόνους. Ε, και ήταν, είχαμε και ένα πολύ ε, ενδιαφέρον ε, άρθρο σχετικά με το, πώς αλλάζουν τα πράγματα σχετικά και με το πώς οι τράπεζες ε, δεν αναλαμβάνουν μακροπρόθεσμη προσέγγιση σε σχέση με τις αποδοχές και με τις πολιτικές πρόσληψεις. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε έχουμε εδώ πολιτιστικά στοιχεία που πρέπει να αλλάξουν γιατί τα συστήματα τα χρηματοπιστωτικά είναι αλληλοσυνδεόμενα και έχουμε και τους κινδύνους στο ιστορικό του συστήματος που πρέπει να ελαχιστοποιηθούν έτσι ώστε όλοι να μπορούν να αναλάβουν τις δεσμεύσεις τους. Ε, αν δείτε την επιχείρηση στη Σκωτία, την RBA, τότε ψήφισαν για την εξαγορά της ε, ΑΜΡΟ μόνο για να ανακαλύψουν ε, οι μέτοχοι στη συνέχεια ότι ήταν υποκατάρρευση η τράπεζα και έπρεπε να συμμετάσχει η κυβέρνηση για να τη διασώσει. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ ε, αν ε, δεν είχαμε σώσει εμείς ε, την τράπεζα θα είχε καταρρεύσει και το σύστημά μας και στη Σκωτία δεν έχουμε πλέον τραπεζικό τομέα Μπορείτε να μιλάτε για μοντέλο οτιδήποτε, αλλά αυτά συμβαίνουν. Έτσι λοιπόν, η εταιρική διακυβέρνηση είναι πάρα πολύ σημαντική και έχει και πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα ο φορολογούμενος. Βλέπετε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα με την οικονομική κρίση, αλλά περαιτέρω στο σημείο 7 αναφέρεται ο κύριος Κάρας ε, ε, ε στην ε, βελτίωση Διακυβέρνηση ε, εδώ σε σχέση με του τιμικού επενδυτέ ε, για να υπάρχει ένα διεθνή κώδικα ορθή πρακτική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Να σκεφτώ τι σκέφτεστε για την ε, ισότητα των δύο φύλων και την ισορροπία των φύλων στα διοικητικά συμβούλια. Σε διοικητικά συμβούλια των τραπεζών υπάρχουν πάρα πολύ λίγε γυναίκε ε, και υπάρχει μια συζήτηση υποχρεωτική συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Θα ήθελα να ρωτήσω του συναδέλφου τι σκέφτονται και για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Αρκετά είπα, σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχουμε πρόβλημα με το χρόνο, γιατί έχουμε καθυστερήσει κατά μισή ώρα. Έτσι λοιπόν, ε, να ζητήσω από τους επόμενους να είναι σύντομοι, γιατί έχουμε δύο ακόμα θέματα. Ο κύριος Φόξ. Ε, thank um, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρετε ότι είμαι εισηγητής για την, ε, στην Επιτροπή ΕΚΟΝ Οικονομικών Υποθέσεων για την ε, έκθεση αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν καταρχάς τον κύριο Κάρας για την γνωμοδότησή του, καθώς επίσης και τους άλλους συναδέλφου για τις δικέ τους παρεμβάσεις. Κύριε Ντιγιό, νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό που είπατε. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε τον φορολογούμενο. Γιατί αν μια εταιρεία πτωχεύσει, τότε απολύονται πάρα πολλοί υπάλληλοι, αλλά δεν υποφέρει ο φορολογούμενο. Ο λόγο όμω για τον οποίο οι χρηματοστατικοί οργανισμοί αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία, ο λόγο για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικέ κυβερνήσει ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη διακυβέρνησή του, είναι γιατί όταν πτωχεύουν οι οργανισμοί αυτοί, το λογαριασμό τον πληρώνει ο φορολογούμενο. Και σε μια εποχή πάρα πολύ σημαντικών δημοσιονομικών περικοπών σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια τέτοια λοιπόν δυσχερή οικονομική περίοδο, οι φορολογούμενοι βλέπουν τα μπόνους των τραπεζιτών και διερωτούνται για ποιο λόγο τα δικά μας τα χρήματα χρησιμεύουν για τη διάσωση των οργανισμών αυτών τη στιγμή που οι δικοί μας οι μισθοί, οι δικές μας οι αποδοχές περικόπτονται. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα αυτό γιατί χρησιμοποιούμε εδώ τα χρήματα των φορολογουμένων για, μια, για ένα συγκεκριμένο τομέα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν τομεί οι οποίοι κατέρευσαν στο παρελθόν, όπω για παράδειγμα ο τομέα τη μεταλλορυχία. Αν θέλουμε αυτή τη στιγμή να διασώσουμε το χρηματοπιστωτικό τομέα, τότε θα πρέπει η δικιά του συμπεριφορά να είναι άκρο υπεύθυνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φόξ. Να δώσω τώρα το λόγο στην Επιτροπή, στον κύριο Έρκιν από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΚΤ. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Ευχαριστώ πολύ για τα πολύτιμα σχόλιά σας. Αναφέρθηκε ότι μπορεί να είναι πολύ αγρά γιατί πολλά κρατημέλη έχουν ήδη αναλάβει κάποιες πολύτιμες δράσεις όπως αναφέρατε, πρέπει να δούμε αν ορισμένε ε, δράσει θα οδηγήσουν σε δραστική αλλαγή συμπεριφορά. Αυτό θα χρειαστεί χρόνο. Γι' αυτό ξεκινήσαμε μια δεύτερη διαδικασία πράσινη βίβλου για να συζητήσουμε εις βάθος ε, αυτά τα θέματα τα οποία αναφέρατε κι εσείς και είναι πολύ ενδιαφέροντα και επίσης ό,τι αφορά και τη σύνθεση των συμβουλίων, των διοικητικών συμβουλίων και την ισορροπία των φίλων στη συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια. Σε αυτή τη δεύτερη πράσινη βίβλο επίσης θα ασχοληθούμε με τη δέσμευση των ε, μετόχων γιατί με δηλώθηκε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε κίνητρα για να μετακινηθούμε από τη βραχυπρόθεσμη σε μακροπρόθεσμη προοπτική. Σε ό,τι αφορά την έκθεση αυτή, είμαστε στη διαδικασία της κατάρτισης. Δεν ε, είναι αργά. Όλα τα πολύτιμα σχολιά σας μπορεί να ληφθούν υπόψη ακόμη και σκοπεύουμε να εκπονήσουμε ένα κείμενο ιδιαίτερα σημαντικό μέχρι τον Ιούνιο. Ευχαριστώ την Κομισιόν για τη συνσφορά της. Τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Κάρας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους ε, για τα πρόσθετα σχόλια και για την υποστήριξή τους. Πρέπει να έχουμε μια πιο δεσμευτική διατύπωση από ό,τι άκουσα. Σε ό,τι αφορά τώρα το σημείο 2, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι συμμετέχουν και οι καταναλωτές. Δεν θα ήθελα στην έκθεση αυτή να ζητήσω νέα ανάλυση. Η ανάλυση των αιτίων της κρίσης έχει γίνει σε πολλές εκθέσεις από πολλές επιτροπές. Δεν έχει νόημα να πω τώρα τι είναι πολύ αργά. Το θέμα είναι να υποβάλουμε τις προτάσεις μας σε σχέση με την πράσινη βίβλο που τώρα έχει υποβληθεί. Μας ενδιαφέρουν τα διοικητικά συμβούλια, οι καταναλωτές και όσον αφορά τα μπόνους ε, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπήρχαν στα CRT και είχαμε σχετικές εξελίξεις στα κράτη-μέλη. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω. Περιμένω τις ε, τροπολογίες σας και θα παρακαλούσα να μου δώσετε τη δυνατότητα να προσπαθήσω να τις συνδυάσω ώστε να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε και να διευρύνουμε τα σημεία που έχουμε εδώ, να μην όμως ε, ε, έχουμε μια εναλλακτική πρόταση σε σχέση με την ε, επί έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάρας. Εγώ θέλω να αναφερθώ στις προθεσμίες. Ε, Σα τις είχα αναφέρει και των 9 ε, Φεβρουαρίου για τις τροπολογίες, στις 12 εξέταση τροπολογιών, 28 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή 28 Φεβρουαρίου, στην ΕΚΟΝ 16 Μαρτίου, ψηφοφορία στην Λομέλεια, ε, τον Απρίλιο του 2011. Συμφωνείτε με αυτό το χρονοδιάγραμμα? Okay. Ωραία. Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο φάκελο που είναι το μέλλον των ε, κοινωνικών υπηρεσιών κοινή ωφέλεια. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Merci, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή για το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος αποτελεί πόρισμα ενός μεγάλου συντονισμού που έγινε με όλους τους ενδιαφερόμενους και τους σκιώδεις ηγητές για όλες τις πτυχές. Μας ενδιαφέρει να έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος για να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα νομικής φύσης. Βλέπουμε ποιες είναι οι τρεις διαστάσεις, η πολιτική διάσταση, η οικονομική διάσταση και η νομική διάσταση των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Θέλουμε μέσω των τριών αυτών αρχών της προσβασιμότητας, της καθολικότητας και της ποιότητας να προσεγγίσουμε τις υπηρεσίες αυτές. Είμαι πεισμένος λοιπόν θα καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο στα πλαίσια της ζήτησης αυτής αν η στάση μας είναι ρεαλιστική και αν, όπως είπε και ο Επίτροπος Μπαρνιέ την προηγούμενη εβδομάδα, και θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ε, ποιότητα της ε, συμβολής του. Αν καταφέρουμε δηλαδή να εφαρμόσουμε την πράξη για την ενιαία αγορά και αν καταφέρουμε μέσω αυτής να δημιουργήσουμε μία νέα ανάκαμψη δυναμική της εσωτερικής αγοράς. Δεν θα ήθελα να φερθώ σε όλα τα σημεία τα οποία έχετε αυτή τη στιγμή στην έκθεση. Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε ένα παρατηρητήριο των, των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντο. Θα καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να χρησιμοποιήσουμε κάποιε βέλτιστε και κοινέ πρακτικέ. Όσον αφορά την οικονομική διάσταση, θέλουμε να καταφέρουμε να συντονίσουμε συγκεκριμένου οικονομικού κανόνε καθώ επίση και τι ιδιαιτερότητε των υπηρεσιών αυτών, κυρίω σε συνάρτηση με του νέου τρόπου οικονομική διαχείριση. Υπότιτλοι Επίσης, όσον αφορά τώρα την ε, νομική διάσταση, δεν μπορούμε να επιλύσουμε όλα τα νομικά προβλήματα, αλλά θέλουμε τουλάχιστον να αποσαφηνίσουμε κάποια νομικά προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει, όπως για παράδειγμα η επικαιροποίηση του οδηγού για τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, κυρίως όσον αφορά την ε, κρατική ενίσχυση και θέλουμε να έχουμε μία ρεαλιστική προσέγγιση και αυτό λόγο ζητάμε το από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσουν σε βάθος συγκεκριμένους ε, τομείς, να δούνε δηλαδή στην πράξη πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί η οδηγία για τις ε, κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Να δούμε δηλαδή πώς μπορούν οι υπηρεσίες αυτές να επηρεάζουν τους ε, συμπολίτες μας. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε εδώ πέρα σε επιμέρους κοινωνικές ομάδες, όπως για παράδειγμα οι ηλικιωμένοι. Επίσης λαμβάνουμε εδώ πέρα υπόψη κάποιες παρατηρήσεις που γίνανε στην συνάντηση με τους κοιόδης ηγητές. Ο κύριος Κορέρα νομίζω ότι είχε ανεβερθεί σε αυτό να γίνει μία αναφορά στην πρόταση 25 της πράξης για την ενιαία αγορά. Αυτά είχα να σας πω τώρα για το χρονοδιάγραμμα. 23 Φεβρουαρίου η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Δεν ξέρω αν θέλετε να διατηρήσουμε την προθεσμία αυτή, αν θέλετε να τη φέρουμε πιο νωρί. 22 Μαρτίου θα γίνει η ψηφοφορία. Στην Επιτροπή Απασχόληση προβλέπεται για τις 24 Μαΐου ψηφοφορία και κατά πάση πιθανότητα θα περάσουμε στην Ολομέλεια του Ιουνίου, αλλά δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα για αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα... Πριν ε, να σας δώσω το λόγο, να επαληθεύσουμε δύο λεπτά το χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, για το Μαΐο και τον Ιούνιο έχουμε την αναβολή. Θα το συζητήσουμε στο τέλος στην συνεδρίασης. Τώρα να δώσω το λόγο στους σκιώδες εισηγητής. Κορέα Δεκάμπος καταρχήν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Αμπάντ για αυτό το πολύ σημαντική γνωμοδότηση. Το άρθρο 3 της Συνθήκης τη Λισαβόνας ε, γίνεται λόγο ε, για την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Το άρθρο 14 αναγνωρίζει τις κοινές υπηρεσίες κοινή ωφέλεια ως τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Αντέλου και το πρωτόκολλο 26 μιλά για την ευθύνη των κρατών μελών στο να διαθέτουν αυτές τις υπηρεσίες και η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αναγνωρίζει το δικαίωμα των πολιτών στην πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Έχουμε μία μια ε, ισχυρή νομική βάση, αλλά δεν υπάρχει ακόμη ορισμό των κοινωνικών υπηρεσιών κοινή ωφέλεια και ούτε υπάρχει ε, ασφάλεια δικαίου και αυτό συνεχίζει να προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα και στο 10. Ε, η πολιτική διάσταση των κοινωνικών υπηρεσιών κοινή ωφέλεια στο πλαίσιο τη κρίση είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι δημόσιε υπηρεσίε Μεταξύ αυτών ε, έχουμε τους παιδικούς σταθμούς, την υπηαγωγία, τη στήριξη στην ηλικία ή στους μετανάστες αποτελούν στοιχεία καθημερινής ζωής των πολιτών. Έχουμε εδώ τρία που πρέπει να προσέξουμε την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ισότητα. Και αυτές οι αξίες πρέπει να είναι ισορροπημένες. Ε, πολλές φορές ε, μπορεί, παραδείγματος χάρη, η αποτελεσματικότητα ε, να είναι κατά της ποιότητας. Πρέπει εμείς να πετύχουμε την ισορροπία. Εσείς κυρία Μπάτ κάνετε μία διάγνωση των αναγκαιοτήτων και καλείτε για ισορροπία μεταξύ κοινωνικής και πολιτικής διάστασης. Εγώ θέλω καλό να γίνει, ε, συμφωνώ με το να γίνει μια μελέτη βάθος επί του τομέα και να βρεθούν τρόποι βελτίωσης της αποτελεσματικότητας. Το κύριο Σεμπάτ ε, υποσπίζει τη διάδοση των πληροφοριών στο διαδίκτυο και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου. Είναι σημαντικό να προωθήσουμε αυτά τα δύο μέτρα. Επίσης, ε, είναι σημαντικό να εμπλέξουμε την κοινωνία των πολιτών και τους πολιτικούς ηγέτες σε αυτό ε, το πρόγραμμα προκειμένου να έχουμε μια καθολική ευρωπαϊκή προσέγγιση αυτών των κοινωνικών υπηρεσιών ε, κοινή ωφέλεια λαμβάνοντας υπόψη τους ε, πολίτες, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, γιατί πολλές φορές ε, παραγωνίζονται ε, και Εμεί θα παρουσιάσουμε κάποιες τροπολογίες για να συμπληρώσουμε το κείμενο. Γενικά όμως συμφωνούμε με την προσέγγιση του συναδέλφου Αμπάντ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ομάδα των φιλελευθέρων, κύριο κύριος Μάντερς. Thank you, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος του Σκιώδου Σιγητού, τον οποίο εγώ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή από την πολιτική μου ομάδα. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή, τον κύριο Νταμιάν Αμπάντ, για τη γνωμοδότησή του Ευχαριστούμε επίση για τη συνάντηση τη σχετική που έγινε τον Δεκέμβριο. Θεωρούμε ότι ο στάκτη γνωμοδότη έχει κάνει μια εξαιρετική εργασία. Κάποιε προτάσει όμω θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη. Εξ ονόματο ομάδα Άλντε, ο σκιώδη ηγητή ε, θεωρεί ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες ε, γενικού ενδιαφέροντος ε, θα πρέπει να αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο, αλλά κάποια τμήματά τους θα μπορούν να ρυθμίζονται και σε κοινοτικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα οι απαιτήσει ποιότητας ή οι κανόνες συνταγωνιστικότητας. Κατά αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει ένα ισότιμο πεδίο ε, δραστηριοποίησης όλων των κρατών. Οι ίδιες συνθήκες συνταγωνισμού θα πρέπει να ισχύουν για όλε τις χώρες. Ο συνταγωνισμό είναι κάτι το θετικό και οδηγεί σε μια πιο καλά λειτουργούσα εσωτερική αγορά. Βέβαια όλοι οι φορείς θα πρέπει να τυχαίουν αξιολόγησης προκειμένου σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει καταπάτηση των κανόνων του ανταγωνισμού. Επίσης ο σκιώδης ηγητής της ομάδας μου πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να έχει να κάνει και με τη γενικότερη αξιολόγηση της ποιότητας που υπάρχει για τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Συμφωνούμε ότι θα μπορεί να υπάρχει, να μια ανταλλαγή δεδομένων στο διαδίκτυο υπό, τον, υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Λέει όμως ότι θα μπορούσαν να ανταλλαγούν και ευέλθυνες πρακτικές καθώς επίσης και άλλες ιδέες από την εφαρμογή των υπηρεσιών αυτών που έχουν τα κράτη-μέλη. Ο Σκιώδης ηγητής σας ευχαριστεί για τις παρατηρήσεις αυτές που του δώσετε δυνατότητα να εκφράσει μέσω εμού και προσβλέπει σε επικοδομητική συνεργασία. Ευχαριστώ. Ρούλε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ε, ζητήσω εκ μέρου ε, του σκιώδου εισηγητή μα, τον κύριο Καμφέ. Ε, θα ήθελα να κάνω κάποιε παρατηρήσει. Να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι στα βασικά θέματα. Τα σήματα 1 έω 3 και 5 δεν είναι προβληματικά. Εγώ προβλήματα βλέπω στο 4 και θα ήθελα να κάνω δύο συμπληρωματικέ ερωτήσει. Όσον αφορά την συνθήκη της Λισαβόνας ε, έχουν αλλάξει τα πράγματα και, έχουν, ε, και έχει ενισχυθεί το θέμα των ε, πρωτογενών συνθήκων. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να φαίνεται πιο καθαρά η αλλαγή, η αυτή δηλαδή στο πρωτογενές δίκαιο. Στο σημείο 5 θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αναφέρεστε σε κατευθυντήριες γραμμές. Υπάρχει το εγχειρίδιο για τις ε, δημόσιες αναθέσεις. Ε, το εγχειρίδιο αυτό όμως δεν είναι επικαιροποιημένο. Εάν αναφέρεστε σε αυτό, τότε θα ήθελα να διαγραφεί η ε, αναφορά αυτή. Μάλλον ε, αποθαρρύνουμε όμως ε, τις ε, τοπικές αρχές. Θα θέλαμε ένα νέο εγχειρίδιο. Και αυτό το έχω ζητήσει και στη δική μου έκθεση για, τις, για τα δημόσια έργα, για, τη, για τις δημόσιες συμβάσεις. Η, το εγχειρίδιο αυτό δεν έχει γίνει με βάση την συνθήκη της Λισαβόνας, αναφέρεται στην παλιά νομική βάση. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι η Κομισιόν αυτή τη στιγμή εκπονεί πράσινη βίβλο για τις δημόσιες συμβάσεις. Ίσως θα μπορούσαμε και εδώ να πούμε ότι θα πρέπει να εξεταστεί πιο προσεκτικά ο τομέας και να διαπιστωθεί γιατί υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, οι οποίες κατά τη γνώμη μου δεν είναι δικαιολογημένες. Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά κριτήρια, ε, ε, είναι αυτονόητο να αναφερθούμε ε, στον τρόπο παραγωγής. Ε, όσον αφορά όμως τα κοινωνικά κριτήρια δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και πάντα δημιουργεί προβλήματα όταν ε, οι δήμοι θέλουν προϊόντα fair trade, δικαίου εμπορίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στριντεφιλίδης. Θα ήθελα να ξεκινήσω και εγώ ευχαριστώντας τον εισηγητή και να θίξω τρία σημεία. Πιστεύω ότι πολύ ορθά η γνωμοδότηση θέτει το προσβασιμότητας, της καθολικότητας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών κοινή ωφελία. Ωστόσο πιστεύουμε ότι στα πλαίσια μιας πλήρους ανταγωνιστικής αγοράς οι πιο πάνω στόχοι μου φαίνονται να είναι ανέφικτοι. Στα πλαίσια του ανταγωνισμού οι πάροχοι των υπηρεσιών δεν θα μπορούν να εξασφαλίζουν τις υπηρεσίες για όλους και ταυτόχρονα να διατηρούν τη βιωσιμότητά τους. Άλλωστε γι' αυτό και το κράτος έχει σε αυτές τις υπηρεσίες ένα τόσο σημαντικό ρόλο. Και το δεύτερο σημείο, ε, νομίζω ότι η Κομισιόν δεν παρέχει ασφάλεια δικαίου στις κοινωνικές υπηρεσίες. Προσπαθεί να διαχωρίσει τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος από εκείνες που δεν είναι εμπορικής φύσης και χρηματοδοτούνται κυρίως από τα δημόσια οικονομικά. Το βασικό κριτήριο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι εάν παρέχονται για το δημόσιο συμφέρον και με αυτή την έννοια το συμφέρον των πολιτών που είναι ταγμένες να εξυπηρετούν. Οικονομικού ή μη οικονομικού ενδιαφέροντος είναι ζωτικές για τον πολίτη, ο οποίος υπόκειται σε φορολογία για να μπορεί να τις απολαμβάνει. Και το τρίτο σημείο πιστεύω ότι είναι πολύ αξιόλογη η πρόταση που κάνει ο εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, το οποίο θα πρέπει να μελετήσει μέτρα που να συμβάλλουν στην τοπική αναβάθμιση της ζωής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην εκπρόσωπο της Επιτροπής, την κυρία Μίλλερ. Είναι εδώ. Δεν είναι εδώ η εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ε. Υπάρχει κάποιος άλλος από την Επιτροπή που μπορεί να μιλήσει. Όχι. Τότε να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή για τις τελικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για όλες τις παρατηρήσεις. Σύμφωνο με τον Αντώνιο Κορέα για το ότι η σημασία αυτών των κοινωνικών ε, επιχειρήσεων ε, ε, μπορεί να αποτελούν ατμομηχανής καιρό κρίσης και νομίζω ότι στην παράγραφο 1 μπορούμε να παρουσιάσουμε αυτή τη διάσταση είναι πολύ σημαντική η διάσταση αυτή και έχουμε μια στέρεα νομική δομή και συμφωνώ εδώ με το ότι σήμερα θα πρέπει να ορίσουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες και το πεδίο εφαρμογή τους και την περίμετρό τους αλλά συμφωνώ επίση και με την ιδέα του για το ότι πρέπει να έχουμε ρεαλιστική προσέγγιση και να μελετήσουμε ένα τομέα. Πολλά σχόλια έγιναν και για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τι κοινωνικέ Υπηρεσίε. Καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει αυτή την ιδέα. Πιστεύω ότι θα επέτρεπε να έχουμε αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και το σύνολο των σχεδόν εισηγητών το υπογράμμισαν αυτό. Κύριε Μάνερ, ε, υπενθυμίσατε τη σημασία τη αρχής ε, της επικουρικότητας ε, είπατε ότι ε, σε ορισμένα σημεία είναι εθνική αρμοδιότητα και γι' αυτό υπενθυμίζουμε στην τελευταία παράγραφο αυτή την αρχή της επικουρικότητας και σε ό,τι αφορά το κοινωνό για τον ανταγωνισμό, συμφωνώ, συνάδελφε, αυτή η διάρθρωση μεταξύ ε, των δημόσιων συμβάσεων είναι σημαντική επίσης για το Βασκαλ Κομφέν συμφωνώ ότι υπάρχουν ε, κάποια θέματα που αφορούν άμεσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποιες ερωτήσεις, ε, γιατί αυτός ε, ο οδηγός μας δείχνει κάποια αρνητικά παραδείγματα. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω στη δική μου έκθεση ότι ένας τέτοιος οδηγός οδεύει μπροστά την κατεύθυνση, αλλά πρέπει να το βελτιώσουμε και ίσως να βρούμε και κάποια θετικά παραδείγματα. Αλλά εδώ καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το εξετάσει αυτό το ζήτημα. Τέλος, ε, σε ό,τι αφορά το συνάδελφο από την Κύπρο, από την ΚΟΕ που υπενθύμησε τις τρεις αρχές ε, των κοινωνικών υπηρεσιών και τον ε, κρατικό ρόλο στον προσδορισμό και την σύσταση των υπηρεσιών αυτών. Να έχουμε ένα πρόβλημα ασφαλείας δικαίου σήμερα και αυτό είναι το παράδοξο γιατί ταυτόχρονα έχουμε στοιχεία νομικά, το επενθύμησε ο Αντώνιο, δηλαδή συνθήκη Λισαβόνα έχουμε το άρθρο 3, και το άρθρο 14 για τις κοινωνικές υπηρεσίες, το πρωτόκολλο 26 και τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έχουμε λοιπόν αυτό το πλωστάσιο, το νομικό, αλλά ορισμό ε, και η πραγματική περίμετρος ε, λείπουν και έχουμε και αποκλήσει μεταξύ των κρατών μελών. Εκεί πρέπει να εργαστούμε λοιπόν και ελπίζω ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο θα μας επιτρέψει να πάμε πιο μακριά σε αυτόν τον καθορισμό τη περιμέτρου. Αυτά για τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν και περιμένω να ακούσω και τις δικές σας παρατηρήσεις για το χρονοδιάγραμμα αν υπάρχουν εξελίξεις γιατί μπορώ να πω ότι αλλάζουν τα πράγματα, είναι μεταβαλλόμενο το χρονοδιάγραμμα. Ναι, πράγματι θέλω να κλείσω αυτή τη συζήτηση κάνοντας μια αναφορά για το πώς έχει κατάσταση με το χρονοδιάγραμμα. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων 27 Απριλίου, δεύτερη ανταλλαγή απόψεων 30 Νοεμβρίου. Αυτό έχει δηλαδή χώρα τελευταία ημερομηνία που δεν συνέπιπτε με όσα είπα. Είναι η εξέταση της έκθεσης 25-26 σήμερα, 23 Φεβρουαρίου προθεσμία για τις τροπολογίες και εξέταση των τροπολογιών και ψηφοφορία στην ΕΜΚΟ 21 22 Μαρτίου. Μαρτίου, ψηφορία στην έμπλη 24 και 25 Μαΐου και κατόπιν ψηφορία στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Συμφωνείτε και εσείς με αυτό το χρονοδιάγραμμα. Πολύ ωραία. Ωραία. Και θα ξαναδώσω την Προεδρία στο Μάρκο. Ευχαριστούμε πολύ. Είσαι σχεδόν συγγήτρια στην επόμενη γνωμοδότηση, έτσι δεν είναι. Θα περάσουμε λοιπόν τώρα στην εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης για την Επιτροπή Μεταφορών όσον αφορά την Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης ε, Επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συντάκτης γνωμοδότησης είναι ο κύριος Κρόιτσμαν, η κυρία Ρούλε, ε, ο κύριος Μπίλε δεν είναι εδώ, ο κύριος Τρενταφυλλίδης όμως είναι εδώ και η κυρία Γκέπχαρντ επίσης σκιώδης συζητητές. Ας ακούσουμε πρώτα την παρουσίασή σας κύριε Κρόιτσμαν και θα γίνει ένας πρώτος γύρος συζήτησης. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, επομένως ζητώ από όλους να είστε σύντομοι στις παρεμβάσεις σας προκειμένου να καταφέρουμε να σημειώσουμε μια κάποια πρόοδο με την εξέταση αυτού του σχεδίου γνωμοδότησης. Έχετε το λόγο κύριε Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο τουρισμός στην Ευρώπη θα πρέπει να γίνει πιο ορατός λόγω της οικονομικής του σημασίας ε, στην Ευρώπη και ε, η ευρωπαϊκή πολιτική τουρισμού μπορεί έτσι να συμβάλλει. Ε, χρήσιμο θα ήταν να ληφθούν κάποια μέτρα για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη. Θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα, θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμα και ε, να εξεταστούν και όσον αφορά την ε, χρηματοδότησή τους. Ε, ενδιαφέρει ε, να κάνουμε πιο ορατή την ε, πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης σε στενή συνεργασία με άλλα όργανα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το θετικό παράδειγμα, η ε, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης μας δείχνει πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Υπάρχει ανάγκη για περισσότερη πληροφόρηση και μεγαλύτερη εξειδίκευση στον τουριστικό τομέα. Ε, έτσι θα μπορούν οι επιχειρήσεις ε, να αντιμετωπίσουν καλύτερα την ε, αλλαγή στον τομέα της ανταγωνιστικότητας. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού χρειάζεται ε, ε, κατάρτιση των ανθρώπων που εργάζονται στον τομέα διότι ε, συμβάλλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού. Χρειαζόμαστε στατιστικά στοιχεία για, την για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό η ποιότητα και ο όγκος των δεδομένων θα πρέπει να συνεπαγόνται προς τη θέμενη αξία. Θα... Ε, πρέπει να επιδιώξουμε ε, βελτίωση του ευρωπαϊκού τουνισμού. Δυστυχώς τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στα διάφορα κράτη-μέλη δεν ε, είναι ενιαία και επίσης ε, οι απαιτήσει των καταναλωτών διαφέρουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Ε, και γι' αυτό ε, μια, μια προσπάθεια να, το επίπεδο να είναι ενιαίο θα μειώσει το επίπεδο. Θέλουμε λοιπόν κάποια συστήματα βαθμολόγησης ε, και θέλουμε η Ευρώπη να γίνει προορισμός για τουρίστες από τρίτες χώρες. θα ήταν χρήσιμο να εμφανίζονται τα κράτη-μέλη ε, σε ενιαία ιστοσελίδα. Υπάρχουν ε, δομές ε, που θα μπορέσουν να διευκολύνουν ε, την ε, ενιαία διαφημιστική προβολή. Θα πρέπει να στηρίξουμε και να διευρύνουμε τις δομές αυτές. Στην έκθεσή μου περιλαμβάνω κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Δυστυχώς ξέρετε ότι υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την έκθεσή μου. Θα Ήθελα όμω ε, πολύ ευχαριστώ να λάβω τι τροπολογίε σα. Αυτά, ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστούμε κύριε Κρότσμαν. Το σημαντικό στην γνωμοδότησή σα είναι ότι επικεντρωθήκατε στα σημεία που αποτελούν αρμοδιότητα τη Επιτροπή μα. Πιστεύω ότι και οι συνάδελφοι θα έχουν να πούνε άλλα πράγματα. Νομίζω ότι έχουμε 15 λεπτά μπροστά μας, πάει λίγο μπροστά το ρολόι της αιθούσης. Μπορείτε πάντως να είστε σύντομοι. Η κυρία Κόμη Γκέπχαρτ, ε, θα μιλήσω και εγώ, ο κύριος Τρεντεφυλλίδης στη συνέχεια και θα ακούσουμε αν έχουμε χρόνο την κυρία Αλιουάσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομη και συλλοπτική. Συμφωνώ με το έργο και τις ιδέες του κυρίου Κρόιτσπερκ ε, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή κληρονομιά. Και τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι υποστηρίζω την αναγνώριση των διπλωμάτων και των προσώπων στο τουριστικό τομέα, γιατί πρέπει να υπάρχει πλήρης εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρώτη πτυχή που θέλω να συμπεριλάβω έχει να κάνει με την εναρμόνιση των προτύπων των ξενοδοχείων. Είχα αναφερθεί σε αυτό το θέμα στην ανταλλαγή απόψεων που είχαμε. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε την ίδια ταξινόμηση και ποιότητα των ξενοδοχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρω ότι είναι ψηλό ο στόχο, αλλά είναι σημαντικό. Και αν πιστεύουμε σε μια ενιαία αγορά, πιστεύω ότι αυτή είναι μια οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε. Μια άλλη πτυχή στην οποία θα επικεντρωθώ είναι ο τουρισμός για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες. Όταν δεν υπάρχουν ε, σχετικές δομές σε όλα τα κράτη-μέλη κατάλληλες ε, για ε, την πρόσβαση των ατόμων με ειδικέ ανάγκες και στα ξενοδοχεία. Αυτό πρέπει να το φροντίσουμε. Επίσης θέλω να αναφερθώ στα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το συνδυασμό με το σήμανση ασφαλείας και τη σήμανση ποιότητας στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Έχουμε και το φάκελο του κ. Ε, για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα πρέπει να συσχετιστεί αυτό με τη σήμανση ποιότητα του τουρισμού. πολλά πρακτορία χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να προωθήσουν τα δικά του τουριστικά πακέτα. Έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρχει πολύ πιο ισχυρή προστασία του καταναλωτή και πρέπει να πιστήσουμε σε αυτό την προσοχή μα. Ελπίζω να ήμουν συνοπτική και ευχαριστώ και πάλι τον συγητή και του συγητές. Ευχαριστούμε πολύ που προσθέσατε κάποια περισσότερα σημεία στην έκθεση. Κύριε Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είμαι σκιώδης ε, εισηγητής. Ε, εκπροσωπώ άλλον συνάδελφο που μου έδωσε κάποιες ε, πληροφορίες. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Το πρώτο θέμα που αναφέρθηκε είναι ότι και σε αυτόν τον τομέα στον τουρισμό δηλαδή θα πρέπει να ασχοληθούμε με νέους τρόπους εμπορίου όπως για παράδειγμα το ηλεκτρονικό εμπόριο και όσον αφορά τις προσφορές και όσον αφορά την ε, χρήση του τομέα αυτού. Θα πρέπει να εξετάσουμε και το τι σημαίνουν αυτές οι νέες ε, συνθήκες και ανάγκες ε, και για τους καταναλωτές και για τους ανθρώπους του τομέα. Όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών σε όλους τους τομείς, έχουμε πολλές διαφορετικές οδηγίες όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών. για τις οδικές μεταφορές, για τις αεροπορικές, για τις συνδρομικές. χρήσιμο θα ήταν να συνοψίσουμε τις, τα δικαιώματα αυτά, να υπάρχει μια ενιαία οδηγία ώστε οι επιβάτες να μπορούν να προσανατολιστούν καλύτερα είναι χρήσιμο να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό οριζόντια. Σημαντικό είναι επίσης ε, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των επιβεβαιών σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα, χρειάζονται μηχανισμοί. Και ο συνάδελφος ο κύριος ε, ε, Κρέγ μου είπε ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το το θέμα αυτό. Σημαντικό ε, επίσης ε, είναι όσον αφορά την εφαρμογή της ε, οδηγίας για τις υπηρεσίες. Το θέμα των διοικητικών εργασιών σημαντικό είναι και το θέμα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Ακούμε συνεχώς τι προβλήματα υπάρχουν, ε, ειδικά όσον αφορά τους tour leaders ε, στις διάφορες χώρες, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα. Επίσης, ε, τα πρότυπα ασφαλείας στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικά και θα πρέπει να εξετάσουμε πώς θα προσεγγίσουμε το θέμα. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες Ε, σημαντικός είναι ο ορισμός των διαφόρων ε, προτύπων ε, όπως είπε η κυρία Κόμη, διότι για παράδειγμα ένας Γερμανός όταν πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων έχει κάποιες προσδοκίες, οι οποίε όμω να μην πληρούνται απαραίτητα από ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων σε άλλη χώρα. Θα πρέπει να σκεφτούμε και το θέμα αυτό και στην ε, όλη συζήτηση επειδή θέλουμε να γίνουμε ο, ο βασικός προ, τουριστικός προορισμός ε, κόσμο, του κόσμου θα πρέπει να σκεφτούμε και τις πιο ήπιες μορφές ε, τουρισμού πέρα από, τις, πέρα από τον μαζικό τουρισμό. Πέρα από τον μαζικό τουρισμό, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ, κυρία... Ρούλε. Ευχαριστώ κυρία Ρούλε και εγώ μπορώ να είμαι πολύ σύντομη. Θα είμαι τα βασικά σημεία τα έχει συμπεριλάβει ο εισηγητής ε, και τον ευχαριστώ για αυτό. Έχει ε, υποστηρίξει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής αυτής. Ε, αναφέρεται στη, στα επαγγελματικά προσόντα, το θέμα της πυροπροστασίας και πιστεύω ότι και για, για το θέμα αυτό θα λάβετε πολλές τροπολογίες και επικροτώ και το θέμα Τη εξάλληψη των ε, προσκομμάτων και τη ε, πρόσβαση ε, για του ηλικιωμένου. Θα μπορούσε ενδεχομένω να προσθέσει κανεί το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου, του ίντερνετ, αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι έχετε θίξει όλα τα βασικά ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τροταφυλλίδης θα μιλήσει πρώτα και θα κάνω κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Ευχαριστήσω τον κύριο Κρόιτσμαν. Πιστεύουμε ότι ορθά η γνωμοδότηση αναγνωρίζει ότι η βάση του σχεδίου δράσης για τον τουρισμό πρέπει να ανταποκρίνεται στο χαρακτήρα της περιοχής για την οποία γίνεται και να αντιμετωπίζει την ιδιαιτερότητα της περιοχής όσον αφορά κοινωνικά ζητήματα, την εδαφική συνοχή και την προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Άλλωστε, η διαφύλαξη των εθνικών ιδιαιτεροτήτων εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει και στη βελτίωση τη συνοχή, αλλά παράλληλα προωθεί και τη διαφορετικότητα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να θίξω είναι ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ε, σημαντική η διαφύλαξη της βιωσιμότητας του τουριστικού προϊόντος με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τον πυρήνα των ξενοδοχειακών παροχών. Άρα και η χρηματοδότηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την στήριξη αυτών των επιχειρήσεων και την παροχή κινήτρων για ανάπτυξη περαιτέρω μονάδων οικογενειακού χαρακτήρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην ασφάλεια και τα δικαιώματα τόσο των τουριστών αλλά όσο και των εργαζομένων στον τομέα. Ευχαριστώ. Να κάνω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Είναι πολύ ενθαρρυντικά αυτά τα οποία ακούστηκαν και πιστεύω θα καταφέρουμε να συμβάλλουμε κι εμείς. Είναι κάπως απογοητευτικό το ότι η έκθεση της ε, Επιτροπής ασχολείται με, τις, ε, με την οδηγία για, την υπηρεσία, τις υπηρεσίες με έναν τρόπο ιδιαίτερα ελαφρύ θα έλεγα. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να λέγεται πόσο πολύ μπορεί να επηρεάσει και τον τομέα του τουρισμού, ότι υπάρχει μία αλληλοσυμπληρωματικότητα αν θέλετε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να το πούμε αυτό τουλάχιστον προς την Επιτροπή ε, Μεταφορών και Τουρισμού. Για κάποια συγκεκριμένα σημεία, η κυρία Γκέπχαρτ αναφέρθηκε στους οδηγούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε στο βιβλίο το οποίο έχει εκδώσει για την πράξη της εσωτερικής αγοράς ότι θα πρέπει να διευθετηθεί το ζήτημά τους και ότι θα μπορούσε να υπάρχει ακόμα και μια επαγγελματική κάρτα για τους τουριστικούς αυτούς οδηγούς. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να αναφερθούμε περισσότερο στο ζήτημα της ασφάλειας και το ζήτημα της ταξινόμησης των ε, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να τονιστεί και επίσης να αναφερθούμε και στην ασφάλεια των προϊόντων που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα αυτά θα πληρούν τις ε, ε, τα απαραίτητα πρότυπα ασφάλειας. Επίσης, θα μπορούσαμε να συνδέσουμε την γνωμοδότηση αυτή με, το, με τη δέσμη μέτρων για τα ταξίδια την οδηγία για τα ταξίδια που θα δούμε στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε εδώ πέρα τον Ευρωπαίο καταναλωτή να αγοράζει κατά τρόπο λογικό και να είναι σε θέση να γνωρίζει βέβαια όλες τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που του δίνονται. Δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο από ό,τι βλέπω η κυρία Αλόης ενδεχομένως να πει κάποια πράγματα εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πείτε μας ποια είναι η δική σας άποψη για τη δική μας εργασία. Ε, ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Καταρχήν σας ευχαριστώ για τα θέματα και τα σχόλια που ακούστηκαν. Νομίζω ότι υπήρξαν ε, ήδη πολλές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις ε, για το θέμα της εναρμόνισης ε, και ότι η Πρόεδρος μας έχει δει τοποθετηθεί, η Κομισιόν ακούει προσεκτικά τις ανησυχίες που εκφράζονται αλλά δίνει και προσοχή στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στον λόγο τομέα σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δικαιωμάτων Καταναλωτών μαζί με τους συναδέλφους ε, διερευνούμε κάθε πιθανότητα για το μέλλον. Σε ό,τι αφορά τώρα τα δικαιώματα των επιβατών, πιστεύω ότι ήδη γνωρίζετε ότι γίνεται μια σημαντική προσπάθεια από τη ΓΑΜΑ μεταφορών να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια ε, να γνωρίζουν οι επιβάτες καλύτερα τα δικαιώματά τους. Δηλαδή υπάρχει μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης ε, μέσω του διαδικτύου. Κάτι ακόμα για τα άτομα ανάγκες. Η Κομισιόν έχει κάνει κάποιες μικρές προσπάθειες με τα μέσα που διαθέτει για να υποστηρίξει προγράμματα που έχουν στόχο τα άτομα με ειδικέ ανάγκε. Φυσικά όμω πολλά ακόμη μπορούν να γίνουν. Εκτιμώ τη συνεισφορά της Επιτροπής και ελπίζω ότι βήμα το βήμα και η της Κομισιόν θα μπορούσαν να υλοποιήσουν τις προτάσεις αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, κάποια σχόλια από τον εισηγητή. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι γνωρίζετε το χρονοδιάγραμμα. Έχει συμφωνηθεί με το Προεδρείο. Σας ευχαριστώ πολύ για τα ενθαρρυντικά σας λόγια υποθέτω ότι θα λάβουν τη μορφή τροπολογιών, τα όσα ακούστηκαν. Νομίζω ότι όλα έχουν συζητηθεί. Άκουσα τι έθιξε και ο Μάλ, και περιμένω τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ. Σε δύο μέρες πρέπει να στέλνουν τροπολογίες, πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε γρήγορα και θα έχουμε και τη συζήτηση 28 Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ όλους ε, για το παραγωγικό πρωινό. Να σας υπενθυμίσω ότι θα ξανασυναντηθούμε στις 3 σε αυτή την αίθουσα. Και έχουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα για σας, ε, για τη Στρογγυλή Τράπεζα, για πιο αποτελεσματική και δίκαιη αγορά, για νικής, ε, για τους καταναλωτέ και τι επιχειρήσει. Σα ευχαριστώ.